Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να αρχίσουμε με τις εργασίες μας. Καθίστε παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι έχουμε σχεδόν απαρτία και θα ήταν σκόπιμο να αρχίσουμε και να ακούσουμε από τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, τους οποίους και καλωσορίζουμε σε αυτή την ακρόαση. Ε, λυπάμαι που κάθεστε αρκετά πίσω ή ίσως να κάνουμε ένα διάλειμμα ενδιάμεσα έτσι ώστε να έρθετε λίγο πιο μπροστά. Αλλά σας βλέπουμε πολύ καλά και από εδώ. Και θα ήθελα να σας πω ότι ακουγόμαστε και στο διαδίκτυο. Βλέπετε και τις κάμερες πίσω σας. Να χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σας και θα φαίνεστε και πολύ καλύτερα από κοντά. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες νομίζω, άρα μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε τη δική σας γλώσσα. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες. Χαίρομαι διότι 22 μέλη από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι παρόντα και θα ήθελα να καλωσορίσουμε για πρώτη φορά ορισμένους συναδέλφους από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο και βεβαίως η Νορβηγία, όπως γνωρίζετε, συμμετέχει πλήρως στην εσωτερική αγορά και εφαρμόζει και την οδηγία περί υπηρεσιών. Χαίρομαι λοιπόν διότι ε, θα δείξετε και ορισμένα ζητήματα από τη δική σας οπτική γωνία ως προς την οδηγία. Ο Μισελ Μπαρνιέ, ο υπεύθυνος επίτροπος, ο οποίος εξελέγει, μάλλον εγκρίθηκε το Φεβρουάριο από το Κοινοβούλιο, θα προσέλθει αργότερα και βεβαίως η ε, μεταφορά της οδηγίας είναι δική του ευθύνη, βασική του ευθύνη. Η μεταφορά της οδηγίας περί υπηρεσιών θα σας πει την, ε, τις δικής, τις δικές του, τη δική του προοπτική και οπτική του όλου θέματος και θα δώσουμε και εμείς και input. Θα ήθελα να καλωσορίσω και την Ήπλιν Γκέπχαρτ, η οποία κάθεται δεξιά μου, που ήταν η συγγήτρια για την οδηγία περί Διορίστηκε το 2003 νομίζω. Το ξέρω πολύ καλά γιατί τότε ήμουν σκιώδης και τώρα είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, έχω αυτό το προνόμιο Άρα βλέπω ότι έχουμε επανενωθεί. Θα σου δώσω το λόγο, Εύλην, να μας κάνεις μια εισήγηση, διότι η Εύελιν είχε την ευθύνη να περάσει η οδηγία από το Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρώπη όταν πέρασε, όταν εγκρίθηκε η οδηγία. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας εμπειρίες για την κοινοβουλευτική διαδικασία και τις έξω κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της οδηγίας. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλά κράτη-μέλη και η ενδιάμεση εξέταση ε, καθώς και οι νομοθετικές αλλαγές ισχύουν και θα συνοψιστούν στο τέλος του έτους. Όπως ξέρετε, ε, υπάρχουν και πληροφορίες για τις επιχειρήσεις Ελπίζω να θυγούν αυτά τα ζητήματα και η κυρία Γκέπχαρτ σήμερα το πρωί ορίστηκε η συγγήτρια από την Επιτροπή για μια πρώτη έκθεση περί μεταφοράς οδηγίας. Επειδή θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη, Θα καλέσω τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων να λάβουν το λόγο. Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι θέλετε να λάβετε το λόγο. Επίσης έχετε και δελτία που μπορείτε να μας δώσετε, τα δείχνει ο Πρόεδρος. Προτείνω λοιπόν να καλέσουμε δύο μέλη από τα Εθνικά Κοινοβούλια, καθώς και μέλη της δικής μου Επιτροπής, έτσι ώστε να έχετε δυνατότητα να ακούσετε και τη δική μας άποψη και μετά να προωθήσουμε έναν διάλογο. Και η Ιβλιν Γκέπχαρτ θα ήταν σκόπιμο να μας εξηγήσει τα σημεία κλειδιά που μας απασχολούν, διότι γνωρίζει πολύ καλά τα περιοδηγίας. Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν να μας κάνει μια εισήγηση η κυρία Γκέπχαρτ. Θα τελειώσουμε σε 6.30 Ίσως γίνει και ένα διάλειμμα, εξαρτάται από την έκβαση της συζήτησης. Στο μεταξύ θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ιβλιν Γκέπχαρτ για να κάνει ορισμένα προκαταρκτικά σχόλια και να μας παρουσιάσει την σημερινή ημερήσια διάταξη. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση έτσι ώστε να συζητήσουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες και να δούμε πού είναι, ποιες είναι οι σημαντικές πτυχές, πού υπάρχουν προβλήματα, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Πριν μπούμε στο πρόγραμμα, να αναφέρω έτσι κάποια ιστορικά σημεία για την οδηγία για τις υπηρεσίες υπήρχαν πολλές πτυχές της συζήτησης, ε, τις οποίες θα πρέπει να θυμηθούμε. Καταρχήν, για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κρατημέλια είναι απολύτω σαφές ότι έχουμε μια κοινή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κοινή αγορά στην οποία πάντα θέλουμε να θέτουμε συγκεκριμένε ε, προϋποθέσεις έτσι ώστε να προστατεύονται και οι επιχειρήσει και οι παροχή υπηρεσιών και οι καταναλωτέ να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, να μπορούν να συνάπτουν συμφωνίε εντό τη επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το εγγυηθούμε λοιπόν αυτό και να το προωθήσουμε, μια βασική προπόθεση ήταν πώ θα διαχειριστούμε την οδηγία για τι υπηρεσίε. Πώ μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό ήταν ο λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε η όλη ένταση, ο καυγά. Η αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν σε κάποια κράτη-μέλη, ε, ονομάστηκε ως ε, οδηγία Μπόλκενστάιν, ήταν η απελευθέρωση, η ιδιωτικοποίηση της ε, αγοράς, όπου καταργούνται οι κανόνες και υπήρχε και άλλη μία ομάδα βουλευτών που έλεγαν όχι, δεν γίνεται να γίνει αυτό, πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο, εναλλακτικό. Και εγώ σε αυτή την ομάδα ήμουν και αυτό πρότεινα. Γιατί είπα ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι θα δημιουργήσουμε κάτι που δεν θα είναι αποδεκτό στα κράτη-μέλη από τους πολίτες. Οπότε έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι το άνοιγμα των αγορών θα συμβάδιζε με, την, ε, με το σεβασμό των ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων, των δικαιωμάτων των κατανοητών και γενικώ των δικαιωμάτων των πολιτών. Τώρα εντάξει, προσπαθήσαμε λίγο να τετραγωνίσουμε τον κύκλο εκείνη την περίοδο και χάρη στην συνεργασία και την πολύ θετική στάση που επεδείχθη στο Κοινοβούλιο, καταφέραμε, παρόλο που για πολύ καιρό θεωρούσαμε ότι δεν θα καταλήγαμε στην ευκαιρία λύση, καταλήξαμε σε μια επιτυχή ε, ολοκλήρωση. Και τα κράτη-μέλη συνεργάστηκαν πολύ, γι' αυτό και τα καταφέραμε ως Κοινοβούλιο να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική πρόταση, θετική συμβιβαστική πρόταση, η οποία μπόρεσε τελικά να γίνει αποδεκτή ομόφωνα σχεδόν από τα κράτη-μέλη. Και τότε είπαμε ότι οι υπηρεσ... οι υπηρεσιών μπορούν να κινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει το δίκαιο των κρατών όπως υφίσταται τώρα να γίνεται σεβαστό. Στο βαθμό που το δίκαιο αυτό είναι θετικό και δεν είναι προστατευτικό, δηλαδή δημιουργεί προστατευτικά προσκόμματα. Και αυτό ήταν ένα από τα σημεία το οποίο έτυχε μεγάλη συζήτηση. Και αυτό είναι μάλιστα και το πρώτο σημείο το πρώτα από τα πρώτα ερωτήματα που ετέθησαν τότε. Είπαμε ότι πρέπει το... να εξετάσουμε το δίκαιο των κρατών μελών και να δούμε ποιοι είναι οι κανόνες που μπορούν να γίνουν αποδεκτοί, που είναι ίσως απαραίτητοι για την κοινωνία και πού βρίσκονται αυτοί οι κανόνες οι οποίοι μπορούν να καταργηθούν και που δεν πρέπει πλέον να ισχύουν. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι απαραίτητο να μελετήσουμε καλύτερα, πιο προσεκτικά το δίκαιο των κρατών μελών και να αξιολογήσουμε τα σημεία που πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε να επιτύχουμε το στόχο μας. Τα πρώτα ερωτήματα που είχαν τεθεί τότε σε σχέση με το θέμα αυτό ήταν το πόσο ε, έγινε αυτό σεβαστό στα κράτη-μέλη, πώς διοργανώθηκε και για μένα ως εισηγήτρια τότε ήταν ε, πολύ σημαντικό και ένα άλλο ερώτημα. Κατά πόσο οι συμμετέχοντες τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των, επιχειρήσεων, οι κοινωνικέ ενώσει, σε όλη αυτή τη διαδικασία πώς μπορούν να εμπλακούν. Γιατί μια τέτοια αξιολόγηση της νομοθεσίας είναι πολιτική αξιολόγηση. Και ξέρω, από όσο άκουσα, ότι στα κράτη-μέλη λήφθη σοβαρά αυτή η αξιολόγηση Εντάξει, υπήρξαν και κάποιοι κανόνες οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταργηθούν μέσω της υπηρεσίας, μέχρι μέσω της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί ως ε, ευρωβουλευτές αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι όταν τα κράτη-μέλη ρυθμίζουν ή δημιουργούν ρυθμίσει ή καταργούν κανόνε και μετά μα λένε Α, οι Βρυξέλλε φταίνε που του καταργήσαμε ή Α, οι Βρυξέλλε φταίνε που δημιουργήσαμε νέου κανόνε, παρόλο που αυτοί ήταν άχρηστοι. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική πτυχή που πρέπει να τη συζητήσουμε. Μετά, σε σχέση με το θέμα αυτό, θέλαμε να μάθουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε στον τομέα αυτό και πόσο βοήθησε και στην εφαρμογή όλων αυτών. Γιατί ξέρω ότι για τα κράτη-μέλη δεν ήταν και πολύ απλό να οργανώσουν αυτό το σύστημα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να συζητήσουμε είναι η δημιουργία των, ενιαίων, των μεμονωμένων σημείων επαφή, των μεμονωμένων συνομιλητών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οδηγία των, για τις υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε όντως να επιτύχουμε την, το άνοιγμα των αγορών, της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μα, να μπορούμε να μιλήσουμε με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο για τον ε, συγκεκριμένο στόχο. Ότι δηλαδή θα γίνεται σεβαστό και το εθνικό δίκαιο και αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν τι απαραίτητες πληροφορίες για το πώς έχει η συγκεκριμένη νομοθεσία, πρέπει να τη σέβονται και πρέπει να δουν τι πρέπει να τηρήσουμε, ποιοι είναι οι κανόνε που πρέπει να σεβαστούμε. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο με το οποίο, το, το οποίο προβλέπεται μέσω των μεμονωμένων συνομιλητών και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και διοικητική διευκόλυνση για τις ε, ε, επιχειρήσεις. Γιατί από τη μία χώρα στην άλλη μπορούν πιο εύκολα να κινηθούν και έχουμε την εμπειρία ότι σε πολλά κράτη-μέλη, ή σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, συχνά πρέπει να δούνε ποια είναι τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν, από τη μία υπηρεσία, πρέπει να σταλούν από τη μία υπηρεσία στην άλλη και πολλές φορές συμβαίνει να είναι 20 ε, υπηρεσίε αρμόδιε. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Θέλουμε να υπάρχει ένας συνομιλητής, ένας άνθρωπος απέναντί μας που μπορούν να αποταθούν οι ε, επιχειρήσει ώστε να λάβουν τι απαραίτητε πληροφορίε και να μπορέσουν να συμπληρώσουν και να διεκπαιρεώσουν όλες αυτές τις τυπικότητε χωρί να πρέπει να μετακινηθούν να μπορεί δηλαδή αυτό να γίνεται και μέσω του διαδικτύου. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό και μια μεγάλη διευκόλυνση για, την, για τις επιχειρήσεις. Και, αυτό είναι, και φυσικά είναι σημαντικό να ακούσω από τα κράτη-μέλη με ποιο τρόπο έγινε αυτό, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε, πού υπήρξαν προβλήματα, πού μπορεί να βρήκατε. Όλα αυτά θέλουμε να τα ακούσουμε. Και ένα τελευταίο σημείο που πρότεινα να συζητήσουμε σήμερα, γιατί δεν είναι δυνατόν να τα συζητήσουμε όλα βεβαίω ένα απόγευμα, ξέρατε τι υπάρχει μέσα από την οδηγία για τις υπηρεσίες, είναι το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Γιατί και γι' αυτό υπήρξε συμβαστική πρόταση και δεν είναι πάντα απόλυτα σαφές ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, γιατί αυτό που είχε προταθεί αρχικά, ότι όλες δηλαδή οι υπηρεσίες κοινού οικονομικού συμφέροντος αποκλείονται, αυτό δεν συνέβη, δεν, δεν προχώρησε. Κάναμε λοιπόν εμείς έναν κατάλογο με τις υπηρεσίες κοινού συμφέροντος, γενικού συμφέροντος, που δεν θέλαμε να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι ιδιαίτερε περιπτώσει και έπρεπε να τι δούμε με ιδιαίτερο τρόπο. Και ξέρω ότι και από κάποια κράτη-μέλη επίση υπήρξαν α, τέτοια αιτήματα. Να αποκλειστούν δηλαδή κάποιε κοινωνικέ υπηρεσίε γιατί εκεί δημιουργεί το πρόβλημα. Οπότε θα ήθελα να δω αν υπάρχουν και άλλοι τομείς που να αντιμετωπίσατε προβλήματα και του οποίου θα μπορούσαμε ίσω να συμπεριλάβουμε εδώ στην συζήτησή μα. Αυτά είναι τα τρία θέματα που ήθελα να σα αναφέρω σήμερα. Βεβαίω ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συζήτηση και πρέπει να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η εφαρμογή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για κάτι και κυρίως τους Γάλλους συναδέλφους. Όταν είμαι στη Γαλλία, πάντα ακούω να μιλάτε για την οδηγία Bolkenstein. Δεν είναι οδηγία Bolkenstein αυτή πια. Έτσι όπως είναι η οδηγία, απέχει πολύ από αυτό που είχε προτείνει ο Μπόλκενστάιν τότε. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να μην δηλητηριάσουμε τη συζήτηση και να λέμε συνέχεια το όνομα του α, υπευθύνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρότεινε αυτή την ε, οδηγία, για να μην α, ε, ε, βάλουμε πολύ νερό στην συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή Ευρώπη η οποία να μπορεί να βασίζεται σε μια όσο δυνατόν πιο ευρεία κοινή βάση. Αυτό πρέπει να προσέξουμε και δεν πρέπει μόνο να δούμε τα προβλήματα, αλλά πρέπει να τονίσουμε και τις θετικές πτυχές. Και γι' αυτό θα σας ήμουν ευγνώμων εάν μπορούσατε να μας πείτε και κάποια θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ξέρω ότι υπάρχουν, γιατί φροντίσαμε να υπάρχουν. Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που έχετε καταβάλει και που είσαστε τόσοι πολλοί σήμερα εδώ, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε. Αυτά που προβλέπονται από την Λισαβόνα, να τα ζούμε, να τα νιώθουμε, να, τα, να αποτελούν εμπειρίε μας. Και η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πάντα σημαντική, θέλουμε να τη βελτιώσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιεκτική αυτή παρουσίαση, οπότε θα θέλαμε να ακούσουμε τώρα τη δική σας άποψη. Η πρότασή μου είναι η εξής. Θα διαβάσω τον αριθμό, τον, τα ονόματα που έχω ήδη ε, στον κατάλογο μου, αλλά αν θέλουν και άλλοι να πάρουν το λόγο, παρακαλώ να μου το γνωστοποιήσουν. Μπορείτε να μας κάνετε νόημα είτε σε μένα είτε στη γραμματεία. Μήπως θα μπορούσατε επίσης ε, εντός τριών λεπτών να τοποθετηθείτε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι και πολύ, πολύ ο χρόνος, αλλά έχουμε και πολλά ε, να συζητήσουμε. Ο κατάλογος μου λοιπόν είναι ο εξής. Την κυρία Πότον από την Νορβηγία, την κυρία Φάιπο Κουνίας από την Σουηδία, τον κύριο Άντριου Σφάμπ, την κυρία Γιάνσον από το Σουηδικό Κοινοβούλιο την κυρία Παπαθανάση από την Ελλάδα, τον κύριο Κασόλη από την Ιταλία και τον κύριο Σεύσικ από την Τσεχία και τον κύριο Λεκού. Για την ώρα αυτούς έχω στον κατάλογο των ομιλητών μου. Θα αρχίσουμε από την κυρία Μπότουν από την Νορβηγία. Τρία λεπτά έχει στη διάθεση σας, κυρία Μπότουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω πώς εφαρμόζεται η οδηγία για τις υπηρεσίες στην Νορβηγία. Σε γενικές γραμμές ε, θα ήθελα να σας επενέσω και εσάς και τους συναδέλφους σας ε, γιατί έχετε συμπεριλάβει και τις ε, χώρες ΕΖΕΣ στην σημερινή ακρόαση γιατί δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις χώρες αυτές. Θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί εταίροι ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να πω ότι η συμμετοχή μας ε, δίνει την δυνατότητα καλύτερη συζήτηση στις χώρες μας. Η πολιτική συζήτηση σε σχέση με την οδηγία για τις υπηρεσίες ε, επικεντρώθηκε κυρίως στο κατά πόσο μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό dumping και ή αν θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Οι, τα συνδικάτα ε, είχαν την δυνατότητα να εισακουστούν και, και εκείνα, να υποστηρίξουν την οδηγία των ε, υπηρεσιών, αλλά ζήτησαν να μην παραβιάζει ε, το δίκαιο των εργαζομένων, τα δικαιώματα των εργαζομένων της Νορβηγίας. Ότι δεν επηρεάζει τις συμφωνίες που ήδη υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Ε, διατηρούνται οι αρμοδιότητες ε, σε σχέση, τα, σε σχέση με υπηρεσίες όπως ε, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η εκπαίδευση κλπ. Έγιναν επίσης εννέα αξιολογήσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τα ερωτήματα που ετέθησαν ήταν κατά πόσο η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα είχε ε, κακές συνέπειες για το εθνικό ε, δίκαιο σε σχέση με την εργασία και τη σχέση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού ε, τομέα. Η αξιολόγηση ήταν ότι κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι δεν ήταν κακός ο αντίκτυπος. Στη συνέχεια πέρασε ένα νομοσχέδιο στο Νορβηγικό Κοινοβούλιο που ουσιαστικά μεταγράφει το, το, την, την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο και την ημέρα που εγκρίθηκε ο νόμος ε, άρχισε να ισχύει η οδηγία στο πλαίσιο της Νορβηγίας. Ε, 1η Μαΐου 2010 είναι η, μέρα... ημερομηνία έναρξης ισχύω σε ολόκληρο τον, τον χώρο ΕΖΕΣ, ε, γιατί έχουν καθυστερήσει στην Ισλανδία με την εφαρμογή. Και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Σε γενικές γραμμές... Ε, ενδεχομένως ε, να υπήρχαν κάποια ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης τα οποία τελικά όμως ε, δεν κρίθηκαν ε, σημαντικά, δεν υφίσταται δηλαδή τέτοιο θέμα, ούτε υπάρχει σύγκρουση με το εσωτερικό δίκαιο της Νορβηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπότεν, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Φάιμπολ Κόνιας από την Σουηδία. Η κυρία, συγγνώμη. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στη Σουηδία, η οδηγία για τις υπηρεσίες ε, ευτυχώς μεταφέρθηκε εγκαίρως στο εθνικό δίκαιο. Κάθε Υπουργείο προσπάθησε να διαπιστώσει ποια είναι τα, τα στοιχεία τα οποία πρέπει να καλύψει η οδηγία και προσπαθήσαμε να δούμε τι εναλλακτικές επιλογές είχαμε. Ως προς τις υπηρεσίες προσπαθήσαμε να δούμε ποια ήταν τα πιο σημαντικά στοιχεία. Εντοπίσαμε ορισμένα προβλήματα, κάποια εμπόδια που υπήρχαν, όπως ε, για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εμπόριο, διαπιστώσαμε ότι έπρεπε αρκετά πράγματα να απλοποιήσουμε στο ε, συγκεκριμένο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much indeed. We are... Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί και εμάς μας ενδιαφέρει πολύ. Ο συντονιστής της ομάδας του ΕΛΚ, ο κύριος Φαμπ, έχει το λόγο. Κύριε Φαμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, ε, κύριος είμαι και όχι κυρία. Ε, θέλω να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τους, ε, τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία αυτή που έχουμε σήμερα εδώ, να είναι και η συγγήτρια της τότε οδηγίας, την συνάδελφο Γκέφχαρτ, και από κοινού να συζητήσουμε ποιο είναι το, ποιος ήταν ο στόχος της τότε οδηγίας. Ότι δηλαδή Μόνο με την εγγύηση κάποιων κοινωνικών και την εξασφάλιση των κοινωνικών προτύπων μπορούμε να είμαστε στην εσωτερική αγορά σε θέση να, να, να εκμεταλλευτούμε όλο το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς. Αυτός ο στόχος είναι που μας ενώνει. Εντάξει, σε κάποιε πτυχέ υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αλλά στην πολιτική συμβαίνει το εξή. Όταν λάβει κάποιο την απόφαση, ε, προσπαθεί να, να επιτύχει του στόχου που έχει θέσει. Ο στόχο τη οδηγία είχε να κάνει και με την, ε, η επίτευξη μάλλον του στόχου είχε να κάνει και με την ε, επίτευξη του σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είναι εξαιρετική η ευκαιρία που έχουμε, που είσαστε εδώ και μπορούμε να συζητήσουμε και για την εφαρμογή και για τις δυσκολίες της εφαρμογής και όλης της διαδικασίας. Και πρέπει να σας πω ότι από τη δική μου την χώρα έχω δει ότι υπάρχει μια σειρά διαφόρων τεχνικών δυσκολιών που προκύπτουν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και στην ε, Γερμανία η, αυτή η μεμονωμένη, ε, τα μεμονωμένα σημεία επαφή είναι κάτι καινούριο ε, για τη δική μου τη χώρα και γενικώ για, το, για τα κράτη-μέλη. Γιατί έτσι μπορεί να διευκολυνθεί πάρα πολύ όλη η διοικητική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών. Η εφαρμογή αυτών των φορέων λοιπόν ε, ήταν, έτυχε λίγο διαφορετικής αντιμετώπισης. Σήμερα έχουμε πολλούς α, μεμονωμένους ε, συνομιλητές, οπότε... Στην αρχή, οπότε μάλλον δεν είναι τόσο αποτελεσματικό το, το, το θέμα αυτό όπως το είχαμε σκεφτεί στην αρχή. Από κοινού όμως πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα αυτά άμεσα και αποτελεσματικά έτσι ώστε να μπορέσει η οδηγία έτσι όπως έχει τροποποιηθεί να εφαρμοστεί πλήρως. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σφαπ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, γιατί ενημερώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών που έχω. η κυρία Γιάνσεν από το Σουηδικό Κοινοβούλιο και μετά η κυρία Παπαθανάση από τη Βουλή των Ελλήνων μετά ο κύριος ε, Κασόλη, ο κύριος Εύσικ ε, από το Τσεχικό Κοινοβούλιο, μετά η ε, συντονίστρια των Πρασίνων, ο κύριος ε, Λεκού και ο κύριος Δεκρό. Και ο κύριος Πάσχα επίσης έχει πάρει το, έχει, θα, θα ήθελε να πάρει το λόγο. Υπάρχει κανείς άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο γιατί πρέπει να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών και οι συντονιστές αν θέλουν, ευχαρίστως να λάβουν το λόγο. Η κυρία Γιάνσεν τώρα από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εύελιν Γκέπχαρτ γιατί μας είπε ότι η οδηγία στην τρέχουσα μορφή της έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με το κείμενο από το οποίο είχε ξεκινήσει. Επίσης η κυρία Γκέπχαρτ μας είπε ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί που έχουν την τάση να κατακρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχουν προβλήματα με τις υπηρεσίες. Όλοι έχουν την τάση να λένε ότι ναι, αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες φταίει». Αυτό συμβαίνει συχνά και στο δικό μας το κοινοβούλιο. Εμείς εφαρμόζουμε την οδηγία αυτή, αλλά έχουμε ένα σημείο για το οποίο δεν συμφωνούμε πάντοτε και αφορά την δυνατότητα επαφής ε, διαλόγου με τα συνδικάτα. Επ' αυτού υπήρξαν κάποια προβλήματα ασυμβατότητας και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, μας είπαν ότι δεν θα ήταν πλέον δυνατό να να διατηρήσουμε ε, το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο πολλές φορές ε, αναφέρθηκε στο Σουηδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να επανέλθουμε σε δεύτερο γύρο παρεμβάσεων. Η κυρία Αφροδίτη Παπαθανάση. Η ελληνική πραγματικότητα τη στιγμή αυτή έχει να κάνει με μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για διαρθρωτικές αλλαγές στη χώρα και για μια βελτίωση των, της δημοσιονομικής κατάστασης και στα πλαίσια αυτά η Ελληνική Βουλή ξεκινά με μια σειρά πρωτοβουλίες, μια σειρά νομοθετικές πρωτοβουλίες στις οποίες περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση της παρούσης οδηγίας. Η οδηγία ψηφίζεται σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είχε κατατεθεί στις 16 Τρίτου στην Διαρκή Οικονομική Επιτροπή από ό,τι βλέπουμε και από το διάλογο που έγινε, υπήρχε η αγωνία για το κοινωνικό ντάμπινγκ, τι θα γίνει με την διαδικασία και την προστασία των υπηρεσιών κυρίως υγείας. Έχει γίνει ένα συντονισμένο διάλογο με του κοινωνικού εταίρου και αυτό ο διάλογο πραγματοποιήθηκε και με τοπικά επιμελητήρια και με συλλόγου και με την παρουσία των, ε, ε, των εργατικών και κοινωνικών εταίρων. Ε, προβλέπεται ότι οι τομεακέ και κανονιστικέ διατάξει των αρμοδίων Υπουργείων θα ολοκληρωθούν μετά την ψήφιση του ανωτέρου νόμου, όπω επίση προβλέπεται ότι τα κέντρα ενιαία εξυπηρέτηση θα στηθούν πάνω στο σύστημα των ήδη υπαρχουσών κέντρων εξυπηρέτηση πολιτών με μια, συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σα ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπουζόη. Θα μιλήσω ρουμανικά, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σας πρωτοβουλία, για διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί στο πλαίσιο της ε, Επιτροπής σας είχαμε πολλές φορές τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Είχαμε πολλές φορές ε, τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Μπαρνιέ. Έχουμε και την έκθεση της εφαρμογής την οποία προετοίμασε η κυρία Γκέπχαρτ. Είχαμε λοιπόν πολλές ευκαιρίες να συζητήσουμε για την εφαρμογή της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες. Όμως δεν, έχουμε καταφέρει, δεν είχαμε καταφέρει μέχρι σήμερα να έχουμε διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ε, την άποψή τους για την εφαρμογή των συγκεκριμένων, της συγκεκριμένης οδηγίας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική οδηγία στο πλαίσιο της εφαρμογής της εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για μια νομοθετική πράξη ιδιαίτερου σημαντική, γιατί η νομοθεσία που θα ισχύσει σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει το θετικό αντίκτυπο της μείωσης της γραφειοκρατίας και της άρσης των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται. Όσον αφορά την κατάσταση στην Ρουμανία, θα ακούσετε από τον εκπρόσωπο της Ρουμανικής Γερουσίας ε, πώς έχει η κατάσταση. Ήταν η δεύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφήρμοσε ε, νομοθεσία συγκεκριμένα προσανατολισμένη ε, οριζόντια νομοθεσία για την οδηγία των υπηρεσιών και μπορώ να σας ε, εγγυηθώ ότι θα υπάρξουν και περαιτέρω προσπάθειες για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας. Πολλές προσπάθειες γίνονται και σήμερα για καλύτερη επικοινωνία, μεγαλύτερο διάλογο με όλα τα κοινοβούλια που δεν έχουν προχωρήσει πολύ στην εφαρμογή της οδηγίας και που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εφαρμόσουν την ενιαία θηρίδα. Γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική οδηγία για το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών και θα ήθελα να, ολοκληρώσω λέγοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε σχέση με την εφαρμογή της ε, εν λόγω οδηγίας είναι ένα παράδειγμα. Δείχνουν τα προβλήματα αυτά, τι εμπόδια μπορεί να υπάρχουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι θα έπρεπε να προβληματιστούμε. Ειδικά για νομοθεσίες που είναι δύσκολο να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο, ίσως θα έπρεπε καλύτερα να επιλέγουμε τον κανονισμό και όχι τόσο την οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ίσως αυτό θα το διερευνήσουμε με τους ε, εθνικούς βουλευτές ως προς τη μεταφορά της νομοθεσίας χρησιμοποιώντας ε, ε, το παρόν ως παράδειγμα. Ο κύριος Κασόλη από τη Γερουσία της Ιταλίας, Σεύσικ, από τη γερουσία της ε, Τσεχίας, την κυρία Ρούιλε, εγώ θα μιλήσω εξ ονόματος της ε, δικής μου ομάδας, από το ΕΛΚΑ, από το Πάσχα και τον κύριο Πάλας, από τους Πολωνούς. Και να σας υπενθυμίσω ότι θα θέλαμε μία εμβαθμένη συζήτηση για τα σημεία ενιαίας επαφής, ενιαίας και μοναδικής επαφής, για να δούμε πόσο έχει εφαρμοστεί η οδηγία μέχρι τούδε και πόσοι συμμετείχαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι ότι οι τοπικές αρχές ή περιφερειακές πολλές φορές είναι αυτές που δίνουν αδειοδότηση στους παρόχους και μας εξέπληξε η κατάσταση Σουηδία όταν μεταβήκαμε τον Οκτώβριο πέρσι γιατί μας είπε η Σουηδική Κυβέρνηση για την διαδικασία ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο για να επεξηγήσουν στην τοπική αρχή ότι τα μέτρα δεν θα έπρεπε να οδηγούσαν σε διακρίσεις ως προς τις αδειοδοτήσεις και πώς θα έπρεπε οι εθνικές αρχές να δράσουν ως προς τη διαδικασία αδειοδότησης τοπικών ή εθνικών παρόχων. Ο κύριος Κασόλη. Και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ, διότι μας δίνετε την ευκαιρία να συνεισφέρουμε κι εμείς. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μας για την εργασία μας, διότι μεταφέραμε την οδηγία περί υπηρεσιών με ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις 8 Μαΐου. Ακολουθήσαμε τις αρχές εξουσιοδότησης που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008, έτσι ώστε να υπάρχει προσπελασιμότητα υπηρεσιών και τροποποιήσεις όπως ορίζονται για τις ε, δραστηριότητες αυτές. Γίνεται μια εξοκοινοβουλευτική δραστηριότητα με τα συνδικάτα έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους φορείς για να κατανοήσουν την οδηγία όπως αρμόζει. Υπάρχουν πολλά κρίσιμα σημεία βεβαίως και ένα από αυτά αφορά την προσπελασιμότητα. Ξαναείδαμε τις προαπαιτήσει για την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση, τροποποιώντας όλες τις διαδικασίες που δεν αρμόζουν με την οδηγία. Επίσης, ακολουθούμε μία διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησης με βάση τα δεδομένα του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να έχουμε και μία νομιμοποίηση ex lege όπως αρμόζει. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το νόμο ως βάση δυνάμει της οδηγίας έτσι ώστε να υπάρξει η σωστή διαδικασία αδειοδότησης από τις δημόσιες αρχές. Τουλάχιστον για την Ιταλική ένομη ε, τάξη πρόκειται για μία καινοτομία έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις και να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης με ευελιξία. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη και την διεύρυνση πελασιμότητα σε αυτή τη δραστηριότητα, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόσβαση σε αυτό, σε αυτό, αυτό το τμήμα των παρόχων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Βεβαίως, πολλές φορές υπάρχουν μεγάλα προβλήματα για τους εμπλεκόμενους φορείς για την σωστή μετάβαση. Τα μεταβατικά μέτρα δεν έχουν προβλεφθεί σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή ε, ως προς τη διαμεσολάβηση θα δούμε κατά πόσο ανταποκρινόμαστε στην ικανοποίηση των ε, συμφερόντων του δημόσιου τομέα, διότι ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να μπορέσει να δράσει και σε αυτό το τομέα. Και θα πρέπει να υπάρχει ε, προσπελασιμότητα με βάση και τις ε, τεχνικές προδιαγραφές. Thank you very much. I think your last point is Ευχαριστώ. Το τελευταίο που αναφέρεται ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η πρόσβαση ε, στην αδειοδότηση είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να χρειαστεί να συζητήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, γιατί έχει άμεση σχέση με τη δουλειά μας και έχει να κάνει και με αυτά που είπε ε, η εκπρόσωπος του Σουηδικού Κοινοβουλίου προηγουμένως. Ο κύριος Σέπτσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς της τσεχικής καμπίνας. Πριν από κάποια χρόνια συζητούσαμε αυτό που τότε ήταν γνωστό ως ε, η οδηγία Bolkenstein. Και επειδή περιμέναμε ότι για κάποιες γειτονικέ χώρες αυτή η οδηγία θα ήταν έτσι ένα είδος δίκτυ για να μειωθεί η περίοδος που θα έπρεπε κανείς να περιμένει ώστε να μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα και να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα, μια επιχείρηση δηλαδή. Του χρόνου ή τα προσκόμματα αυτά θα έχουν αρθεί. Και η τσεχική οικονομία αλλά και οι γειτονικέ οικονομίες δεν έχουν υποφέρει και πολύ λόγω αυτής της μεταβατικής περίοδου. Μάλλον ψυχολογικό ήταν περισσότερο παρά οικονομικό το κίνητρο. Ήταν δεκτό για μας να απελευθερώσουμε περισσότερο τους τομείς της οικονομίας μας. Προχωρήσαμε λίγο παραπάνω από αυτά που ζήταγε η ε, ο δικός μας, ε, η δική μας νομοθεσία είναι πιο φιλελεύθερη, πιο ευρεία σε αφορά την απελευθέρωση των υπηρεσιών και έχει, ενέχει πολύ, περισσότερες, ε, πολύ περισσότερους τομείς σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Έχουμε και τέτοια εμπειρία εμεί με τα σημεία επαφής, με τα κέντρα ενίας εξυπηρέτησης. Δύο υπάρχουν στην πρωτεύουσα. Βέβαια, αν υπάρξει μεγαλύτερη προώθηση, εντάξει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ακόμη περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιούνται τώρα. Νομίζω ότι αυτή η φιλελεύθερη άγουσα που έχουμε πάρει είναι ε, ε, θετική, αν δούμε και τις απαντήσεις του πολιτικού κόσμου. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διευθυντήσει τα θέματα αυτά με πιο φιλελεύθερο τρόπο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια τη Τσεχική Προεδρία πριν από κανένα χρόνο έγινε μια μεγάλη διάσκεψη για την εφαρμογή τη οδηγία στην Πράγα και πραγματικά έχει λάβει. Έχουν, έχει δώσει, μάλλον έχουν δώσει πολλές προεδρίες μεγάλη σημασία σε αυτή την οδηγία. Ίσως αυτό να είναι έτσι ένα κίνητρο για να πράξουμε αντιστοίχως και για άλλες ε, οδηγίες. Η κυρία Ρούλε, θα είμαι σύντομη γιατί ήθελα καταρχήν να ακούσω τι έχουν να πούνε οι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων γιατί βασικά τις δικές τους εμπειρίες ήρθαμε να συζητήσουμε εδώ με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ακούστηκαν κάποια σημεία ε, Παρ' όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι η εφαρμογή δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε διάφορε χώρε και ελπίζω να εξακολουθήσει να υπάρχει το ενδιαφέρον ε, και να μπορέσουμε να ακούσουμε και άλλε εμπειρίες από του καλεσμένου μα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεκρού. Merci, monsieur le... Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ο κύριος Λεκού είμαι. Είναι δύσκολο μερικές φορές να προφέρει κανείς ε, τα ονόματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να απαντήσω στην ε, κυρία Γκέπχαρ, την ε, εισηγήτρια που έθεσε το ερώτημα και είπε μάλιστα ότι στη Γαλλία πολλές φορές ε, την ε, ε, αποκαλούμε ακόμη οδηγία Bolkenstein, την, την οδηγία για τις υπηρεσίες. Όχι, σας διαβεβαιώ ότι αυτό δεν ισχύει πλέον, παρά το γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ την, τη γαλλική κοινή γνώμη, ειδικότερα όταν πρόκειτο να εκφράσει την άποψή της η κοινή γνώμη για μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη. Εμείς ε, είχαμε τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε ε, στη Γαλλία όταν ε, είχαμε, είχατε έρθει για να συζητήσουμε ακριβώς στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής. Έχει εξελιχθεί λοιπόν πολύ αυτή η οδηγία και ελπίζουμε ότι ακόμη περισσότερο θα εξελιχθεί με τη συμμετοχή και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι γεγονός ότι είναι βαρύ το καθήκον της μεταγραφής της νομοθεσίας αυτής στην Εθνική Νομοθεσία, γιατί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι πολύ ευρύ. το βαρύ αυτό λοιπόν καθήκον το έχουμε αναλάβει και η κυβέρνηση έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση γιατί υπάρχουν ορισμένα κείμενα τα οποία είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο γίνεται και από το ίδιο το Κοινοβούλιο. Μερικέ φορέ όμω, νόμοι που ψηφίζονται στο Κοινοβούλιο χωρί πρωτοβουλία τη κυβέρνηση, ε, τα προτείνουν οι ίδιοι οι βουλευτέ. Όλο ο κόσμο λοιπόν συμμετέχει προκειμένου να ε, γίνει αυτή η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Παρά το γεγονό ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο εγχείρημα, πολλές φορέ ε, έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Θα γνωρίζετε κι εσείς ε, ότι, ε, να για παράδειγμα ψηφίσαμε το νόμο εξυγχρονισμού της οικονομίας. Ε, ε, έχουμε επίσης έναν άλλο νόμο για τον εξυγχρονισμό της ανάπτυξης του τουρισμού, για τη διευκόλυνση της δραστηριότητας πολίσεων στον τομέα του τουρισμού ή της, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Και θέλω, σας το λέω αυτό για να σας πω ότι καμιά φορά οι τίτλοι των ε, νόμων ε, δείχνουν ακριβώς πόσο ε, μεγάλη εμβέλεια είναι το εγχείρημα. Για παράδειγμα, υπήρχε ένας νόμος για τα νοσοκομεία. Πολύ γενικό και γι' αυτό πολύ δύσκολο. Και κατά τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μία ακόμη νομοθεσία τέτοιου είδους με πρωτοβουλία των βουλευτών για να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι προσπάθειες. Μερικές φορές μάλιστα ε, ακόμη και τα νομικά επαγγέλματα και πολλές φορές ε, μάλιστα έχουμε την ε, ιδιαιτερότητα στη Γαλλία ότι υπάρχει αντίσταση πολλές φορές σε τέτοιου είδου ε, αλλαγές, όμως πρέπει να προχωρήσουμε. Όσον αφορά λοιπόν την ε, ενιαία θηρίδα, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ενιαία θηρίδα ε, που διευκολύνει την ομοθεσία αυτή. Μιλάμε για το κέντρο διαδικασιών που αφορούν τις επιχειρήσεις, δηλαδή και ενημερώνει το κέντρο αυτό και καταχωρεί. Ιδού λοιπόν μια οδηγία η οποία κάποτε με το πρώτο της όνομα μας δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αλλά σήμερα σιγά σιγά θα μπει στα γαλλικά ήθη αλλά παρόλα αυτά δεν σας κρύβω ότι το πεδίο εφαρμογή είναι τόσο μεγάλο που πολλές φορές αναρωτιόμαστε μήπως έχουμε φτάσει στα όρια του λογικού με ένα τόσο ευρύ πεδίο εφαρμογής. Ε, αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Uh, um, Ευχαριστούμε κύριε Λεκού και ίσως ε, μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα της ε, ενιαίας θηρίδας ή των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης, ε, γιατί θεωρείται σημαντικό από πολλούς. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους των άλλων κοινοβουλίων για την τεχνολογία που διαθέτουμε εδώ. Ήμασταν η πρώτη επιτροπή, επιτροπή εσωτερικής αγοράς, που είχαμε μια κοινή τηλεδιάσκεψη με μια επιτροπή σε ένα άλλο κοινοβούλιο, δηλαδή με την Εθνική Εθνοσυνέλευση, τη Γαλλική, την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, όταν μιλήσαμε για την οδηγία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Όχι σε αυτό το κτίριο, σε ένα άλλο, αλλά χρησιμοποίησαμε το, τον ίδιο εξοπλισμό τις ίδιες οθόνες, διερμηνία και ούτω καθεξής. Άρα καλούμε τα εθνικά κοινοβούλια που διαθέτουν τέτοιο εξοπλισμό να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία και να συνεχίσουν να προωθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Assemblée Nationale, μου έγραψε και ο πρόεδρος της Γενικής Εθνοσυνέλευσης και ήταν ιδιαίτερα επιτυχής η τηλεδιάσκεψη. Κύριε Ντεκρόμ, ελπίζω να προέφερα σωστά το όνομά σας από το Βελγικό Κοινοβούλιο. Ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σε όλες τις γλώσσες του τόπου. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την διοργάνωση αυτής της ε, συνάντησης Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι έχουμε εγκρίνει την οριζόντια οδηγία και είμαστε στην διαδικασία έγκρισης της εγκάρσιας οδηγίας και όπως γνωρίζετε είμαστε μια ομοσπονδιακή χώρα και υπάρχουν πολλές πτυχές της οδηγίας που θα πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν από τα περιφερειακά κοινοβούλια. και αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό συζήτηση. Άρα δεν έχουν ε, μεταταχθεί στην εθνική νομοθεσία, αλλά αυτό θα γίνει σε λίγες εβδομάδες. Ως προς την ε, ουσία, ο κύριος Μπόλκενστάιν ήταν προσωπικός μου φίλος και είναι. Το 2002 συνέταξε αυτό το προσχέδιο οδηγίας και στόχος ήταν να προσπαθήσουμε να άρουμε πολλά από τα προσκόμματα στο εμπόριο. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα και να εξεύρουμε ε, τρόπους έτσι ώστε το εμπόριο να συνάδει με τις αρχές του ανταγωνισμού. Αυτό είχε κατά νου τότε και όπως είπατε το όνομα εμένει και έχει επιβιώσει. Αυτό δεν έχει όμως σημασία. Σημασία έχει να δούμε τις επιπτώσεις της οδηγίας ως προς την ευημερία γενικότερα, σε, ως προς τα επίπεδα απασχόλησης και για να άρουμε τα τεχνικά προσκόμματα. Θα πρέπει να πω ότι έχουμε να κάνουμε με μια οδηγία η οποία έχει ευνουχιστεί. Το δεύτερο βασικό σχόλιο είναι ότι ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι οικονομικές πτυχές διέπουν την όλη οδηγία και ως προς τους σιδηροδρόμους, τα ταχυδρομεία διέπονται από τις ίδιες αρχές και έχουμε προβάλει μία νοοτροπία αυτοπροστασίας, η οποία είναι πολύ κοντόθωρη κατά τη δική μου άποψη. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήμουν Υπουργό, στο υπεύθυνο για το δίκτυο σιδηροδρόμων στις μεταφορές η κάθε χώρα έχει τη δική της νομοθεσία στον τομέα των σιδηροδρόμων διότι θεωρεί ότι είναι η πρόσωψη μιας χώρας. Αυτό όμως είναι πολύ αρνητικό, διότι έχω την εντύπωση ότι σε μια κατάσταση παγκοσμιοποίησης, σε μια παγκόσμια οικονομία, όλα αυτά τα προσκόμματα θα πρέπει να αρθούν. Και παρά τις οδηγίες που προσπαθούμε να θέσουμε σε εφαρμογή, πολλές φορές αυτά τα προσκόμματα ισχύουν. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much indeed, Mr. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης έχει μείνει στην, στον καταλογό μου. Ο κύριος Πάνας από τη Ρουμανική Γερουσία και ο κύριος Μπένις από την Πολωνική. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους υπόλοιπους να πάρει το λόγο. Θέλουμε να ακούσουμε όσο, ε, όσο περισσότερες εμπειρίες δικές σας μπορούμε, ε, γιατί εσείς ήσασταν αυτοί που ασχοληθήκατε επί τόπου, πώς ήρθατε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτά που υπόθηκαν. Κάντε μας ένα νόημα, ένα ανέβημα για να σας δώσουμε το λόγο. Να δώσουμε το λόγο καταρχήν στον κύριο Τρετοφυλλίδη και μετά στον κύριο Πασκάλ και στον κύριο Μπάνας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την ε, ευκαιρία για να έχουμε αυτό το feedback από τις Εθνικές ε, Βουλές, από τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ επίσης ε, για την διοργάνωση του, του hearing, αλλά ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τις αλλαγές που η συνάδελφος Κέμπαρντ έχει επιτύχει στην οδηγία και έτσι με χαρά θα την ονομάζω εγώ τουλάχιστον οδηγία Γκέμπαρντ αντί οδηγία Μπόλκεστάιν. ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν πάρα πολλοί ε, πολύπλοκες ε, στην οδηγία αυτή που εμποδίζουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με την εφαρμογή της, αν κρίνει κάποιος από τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Φεβρουαρίου της Επιτροπής. Εκεί αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι 13 κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει τον νόμο πλαίσιο με τον οποίο η οδηγία γίνεται μέρος της εσωτερικής τους νομοθεσίας, αλλά σε άλλα ε, δέκα κράτη-μέλη η οδηγία βρίσκεται ενώπιον των Εθνικών Κοινοβουλίων ακόμα, ενώ σε δύο κράτη-μέλη η νομοθετική επεξεργασία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ε, φαίνεται ότι αυτές οι δυσκολίες αναγκάζουν τα μέλη να ε, ε, προβληματιστούν ακόμα περισσότερο και ήθελα να τονίσω ότι για μας δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός να πιέσουμε τα κράτη-μέλη, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να πιέσει τα κράτη-μέλη για την τάχιστη εφαρμογή της οδηγίας και όλων αυτών των πολύπλοκων προνοιών της, αν τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα ακόμα. Ε, μια βεβαιασμένη εφαρμογή μπορεί να προσθέσει στα προβλήματα που ούτως ή άλλως αναμένεται να υπάρξουν. Έτσι θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχουμε ακόμα λίγη υπομονή. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, θα δούμε ε, αν θα καταφέρουμε να συζητήσουμε για τα αποτελέσματα. Ο κύριος Πασκάλ από την Ορμανική Γερουσία. Ε, Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους ευρωβουλευτές και βουλευτές που είναι παρόντες στην ε, Ρουμανία στα πλαίσια της προετοιμασίας ολοκλήρωσης προσπαθούσαμε, προσπαθήσαμε να άρουμε τα προσκόμματα που υπάρχουν και στο γλωσσικό τομέα και, στο, και γενικότερα. Γιατί αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να δούμε την διαδικασία αδειοδότησης ως προς τις νέες ευκαιρίες που προβάλλονται και μέσα στα πλαίσια της απλούστευσης έτσι ώστε να μειώσουμε τον αριθμό αιτήσεων και να πλουστεύσουμε και την τεκμηρίωση για το κόστος αδειοδότησης. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες σε σχέση με άλλες χώρες, διότι σημασία έχουν και οι διασυνοριακές υπηρεσίες, θα θέλαμε να δούμε πώς έχει η διαδικασία αδειοδότηση σε άλλα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Βεβαίως, πολλές φορές υπάρχουν θέματα γενικού εθνικού συμφέροντος Τέλος, η διαδικασία ε, αμοιβαία αξιολόγησης θα μας οδηγήσει σε συμπεράσματα μέσα στα πλαίσια της ενδεχόμενης εναρμόνισης για να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ. Uh, thank um, Ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Μπανιάς από την Πολωνική Γερουσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, η οδηγία για τις έχει μεταφερθεί στο πολωνικό δίκαιο ήδη με νομοσχέδιο από το Μάρτιο του 2010 για την παροχή υπηρεσιών στην Πολωνία που καθορίζει συγκεκριμένες, κανόνε κανόνες και αλλάζει 27 εφαρμοστικές πράξεις. Εγκρίθηκε απόλυτα και από τα δύο ε, και από, την, ε, και από, τις, ε, και από το κάτω και το άνω κοινοβούλιο και ο πρόεδρος Κατσίνσκι είχε υπογράψει το νομοσχέδιο που άρχισε να ισχύει στις 10 Απριλίου του 2010. Συμβολική ημερομηνία για μας, ξέρετε γιατί. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε ό,τι αφορά κυρίως την Πολωνία. Σε κάποιες ε, επαναστατικές διατάξεις για την δι διοικητική, τα διοικητικά, δηλαδή τη διοικητική απλούστευση. Έχουμε και την ε, συμφωνία που έχει συναυθεί, δηλαδή υπάρξει ένα, περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς απάντηση, ο ετών λαμβάνει αυτόματα άδεια για να κάνει τις ε, ε, επιχειρήσεις του. για την απόδοση άδεια παρατείνεται μόνο μία φορά η προθεσμία. Αυτό είναι αρκετά επαναστατικό για τα πολωνικά δεδομένα. Και πρέπει να παρακολουθούμε πολύ λεπτομερώς τους νόμους μας, γιατί αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ καινούργιο για, τους, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Αυτά ήθελα απλώς να σας πω. Σας ευχαριστώ. Uh, well, thank you very much indeed, uh, uh, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Μπανιάς. Γνωρίζουμε την τραγωδία στη χώρα σας. Ε, έχετε τα συλληπιτήρια όλων μας. Κάποιο σχόλιο να κάνω κι εγώ. Γιατί έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος των ε, ομιλητών και πρέπει να δώσω το λόγο και στην Εύελιν. Ίσως στην επόμενη, στο, στην επόμενη ανταλλαγή απόψε να μπορέσουμε να μπούμε λίγο στη λεπτομέρεια του πράγματος. Από τη δική μας την πλευρά, νομίζω ότι ένα από τα πιο, μία από τις πιο βασικές πτυχές αυτής της οδηγίας είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε αυτή την γενική διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης. Καλό θα ήταν ε, στις υπόλοιπες παρεμβάσεις σας που ίσως κάνετε, να μας πείτε αν αυτό είναι διοικητικό στη χώρα σας, πόσο έχει προχωρήσει, γιατί όλη αυτή η ιδέα του ότι όλες οι χώρες ή σχεδόν όλες οι χώρες κάνουν μια ολομέλεια για να συγκρίνουν ε, εμπειρίες, για να μελετήσουν ε, τα, το τι συμβαίνει είναι εντάξει, ένα εγχείρημα αρκετά περίπλοκο αν δείτε τις, ε, το τι λέει το Συμβούλιο Μιλούμε για πάνω από 19.000 ε, διατάξεις, ε, τις οποίες πρέπει να εξετάσουν τα 27 κρατη ε, Υπάρχει λοιπόν μεγάλη δέσμευση, έτσι, εμπλοκή, ανταλλαγή εμπειριών. Αυτό είναι κάτι καινούριο όμως σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και βεβαίως θα θέλαμε να δούμε ποιες είναι οι δικές σας απόψεις για μια τέτοια πολιτική διαδικασία γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς. Και πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, για να δούμε ποια κομμάτια της νομοθεσίας ίσως καθυστερούν, επιβραδύνουν την όλη, το όλο μας εγχείρημα. Βεβαίω, τα κρατημέλη δικαίω θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των, πελατών, των πολιτών του ό,τι αφορά την δημοσία υγεία, να τηρούνται ε, τα, κριτήρια που έχουν μπει στην οδηγία. Αυτό από μόνο του είναι πραγματικά μια νέα ε, αξιοθαύμαστη διαδικασία και γίνεται κυρίω σε διοικητικό επίπεδο προς το παρόν. Οπότε θα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσε οι δικέ σα απόψει για τα θέματα που απορρέουν από όλο αυτό. Και δεύτερο, αυτό που είπε ο κ. Μπανιάς για τις διοικητικές διαδικασίες και το γεγονό ότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε από τη δουλειά που έχει γίνει, που οδήγησε στην εκπόνηση της οδηγίας, ότι ένα από τα αντικίνητρα ε, μια επιχείρηση να πάει να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα είναι ότι έκανε ανέτηση για άδεια και δεν έλαβαν ποτέ απάντηση για άδεια Και μετά πήγαιναν και έκαναν κάτι άλλο ή πήγαιναν σε κάποια άλλη χώρα αυτή η δυνατότητα ή η ανικανότητα καλύτερα απάντησης ήταν ένα από τα προσκόμματα. Και χαίρομαι που το έθιξε ο κύριος Μπάνος αυτό, γιατί νομίζω ότι οι επιχειρήσεις στην Πολωνία και οι πολίτες της Πολωνίας κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, θα απεφοληθούν τώρα, γιατί θα απαντάτε μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το αίτημά τους. Και ένα άλλο που θέλω να δείξω και που προκύπτει από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει ήδη από σήμερα το πρωί με κάποιους από τους συναδέλφους από την Βρετανική κυβέρνηση είναι ότι αυτή η οδηγία οδηγεί σε απλούστευση του επιχειρησιακού, επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε όλες τις ε, χώρες. Αυτή είναι η δική μου θεωρία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θα μου το πείτε. Αλλά αυτό το να μην απαντά κανεί σε αιτήματα δείχνει ότι όντω τώρα ε, βελτιώνεται η κατάσταση. Και αυτό έχει παρατηρηθεί και σε, για τι πολωνικέ επιχειρήσει, όχι μόνο σε περίπτωση που θέλουν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα, αλλά και εντό τη χώρα του. Οπότε όλο αυτό, όλα αυτά τα ωφέλη προκύπτουν από αυτή την γενική διαδικασία ε, εσωτερική ανάλυση τη νομοθεσία. Βλέπω ότι κάποιο Κάποιος θέλει να πάρει το λόγο εκεί πίσω. Όχι, κάποιος σήκωσε το χέρι. Όχι, δεν θέλετε να μιλήσετε. Εντάξει. Ωραία, αυτές λοιπόν οι παρατηρήσεις οι δικές μου. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε σχόλια. Αν δηλαδή και στην πράξη όντως έχετε παρατηρήσει αυτό που σας λέω εγώ θεωρητικά, ε, αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, η Εύελιν να κάνει ίσως κάποια καταληκτικά σχόλια και μετά να περάσουμε στο επόμενο τμήμα. Yeah, ε, Ευχαριστώ. Ε, με βάζετε σε δύσκολη θέση, Πρόεδρε, γιατί μιλήσατε για ένα, προ... για ένα θέμα το οποίο δεν είχαμε καν προβλέψει να συζητήσουμε. Αλλά εντάξει, μπορώ να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Αυτή δηλαδή την αμοιβαία ε, αξιολόγηση που προβλέπετε. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους εδώ τους συμμετέχοντες ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση είχε αρνηθεί αυτή την αμοιβαία ε, αξιολόγηση. Την είχε διαγράψει σχεδόν ομόφωνα με τις ψήφους όλων των ομάδων, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ γραφειοκρατική η διαδικασία, πολύ γραφειοκρατική η ιστορία και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη ήταν αυτοί που ήθελαν οπωσδήποτε να υπάρχει αυτή η αξιολόγηση. Και στη δεύτερη ανάγνωση είπαμε εντάξει, αν το θέλουν τα κράτη-μέλη, ας το πράξουν. Θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, οπότε φυσικά και εμείς δεν θέλαμε να τους εμποδίσουμε. Αλλά να μην καταλήξουμε στο ότι το Κοινοβούλιο ε, εγκαταστάθηκε αυτό το γραφειοκρατικό τέρας. Η Πολωνία πρέπει να αξιολογήσει τι γίνεται στα υπόλοιπα 26 ε, κρατημέλη και τα υπόλοιπα 26 κρατημέλη επίσης. Μιλάμε δηλαδή για πολλή δουλειά. Και αυτό όλο υπό την αιγίδα του, της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. με φαίνεται σε δύσκολη θέση, Πρόεδρε, που πρέπει να τα θυμίσω, τα που θυμίσω τα γεγονότα. Τώρα, αυτό που άκουσα από τις απαντήσεις και που είναι σημαντικό για μένα και θα ήθελα ίσως για κάποιες ακόμη πληροφορίες για το πόσο εντατικά τα κοινοβούλια ασχολήθηκαν με αυτή την ε, αξιολόγηση, την επαλήθευση των δικαιωμάτων, των, των νομοθεσιών που έπρεπε να αλλάξουν, ε, των πράξεων που έπρεπε να προσαρμοστούν, δηλαδή το πολιτικό επίπεδο πόσο ασχολήθηκε με όλη αυτή την ιστορία, όχι μόνο οι τεχνοκράτες. Σίγουρα οι δημόσιοι υπάλληλοι έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους, δεν ε, θέλω να τους δείξω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις οι οποίες είναι υψηλά ε, πολιτικές και καλό θα ήταν να ακούσουμε πόσο εντατικά έχει εμπλακεί σε όλη αυτή τη διαδικασία το πολιτικό επίπεδο. Ξέρω ότι σε κάποια κράτη-μέλη αυτό έχει γίνει ε, στεναρά, ξέρω σε κάποια κράτη-μέλη άλλα. Ε, είναι λίγο πιο χαλαρέ οι συνθήκε, ε, έχει αφαιθεί στα χέρια των υπαλλήλων. Και θα ήθελα να μου πείτε λίγα πράγματα παραπάνω γι' αυτό. Δεύτερον, πολύ ενδιαφέρον που ακούστηκε είναι αυτή, αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις Πώς δηλαδή διαχειριστήκατε όλη αυτή την νομοθεσία. Σε ένα κράτος μέλος είναι, γίνεται με οριζόντιο τρόπο. Μα είπε ο συνάδελφο από την ε, Ιταλία α πούμε. Καλό θα ήταν ναι, ο κύριο Κασόλη, αν μπορούσε, να μας πει πώς τα καταφέρατε στην Ιταλία. Και ένα άλλο παράδειγμα, αυτά που είπε ο συνάδελφος από τη Γαλλία, που είναι πολύ ειδική η νομοθεσία που προβλέφθηκε έτσι, να σας δείξω δύο αντικρουόμενα πούμε, παραδείγματα, τα οποία όμως λειτουργήσαν εξίσου. Να μας πείτε και εσεί ποιο ήταν, ποιος, ποια ήταν η προσέγγιση σας. Καλό θα ήταν να ακούσουμε τι συγκεκριμένα κάνατε, τι αλλάξατε, πώς, τι συνέπειε είχε όλο αυτό σε ό,τι αφορά την νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λίγο περισσότερες πληροφορίες. Βέβαια, ε, ευχαρίστω και γραπτό είμαι email να ανταλλάξουμε αυτέ τι ε, πληροφορίε, να ρωτήσω, να θέσω εγώ τα ερωτήματά μου και αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι συνάδελφοι ασχολήθηκαν πολύ περισσότερο με το δεύτερο σημείο για τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην οδηγία για τις υπηρεσίες, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά των κρατών μελών. Γι' αυτό πραγματικά περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσω τι θα μας πούνε στο δεύτερο γύρο για το συγκεκριμένο αυτό σημείο οι συνάδελφοι. Σα uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύλην. Έχουμε περιορισμό χρόνου. Έχουμε βεβαίως χρόνο ομιλίας και γι' αυτό νομίζω ότι θα εγκαταλείψουμε το όριο των τριών λεπτών, γιατί έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και θα έπρεπε να προωθήσουμε έναν διάλογο. Ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για τα κέντρα ενίας εξυπηρέτησης ή τις ενιαίες θηρίδες. Άμα θέλετε λοιπόν να αναφερθείτε, να σε άλλα σημεία στα οποία προαναφέρθηκε κάποιος, όλα τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα κυρία Μπότν ήθελε να ε, μιλήσει για τα κέντρα ενίας εξυπηρέτησης, αλλά όποιος άλλο θέλει μπορεί να συνεισφέρει. Απλώς να μας ε, αναφέρετε, αν θέλετε το λόγο, κυρία Μπότον θα αρχίσει τη συζήτηση και οποιοδήποτε άλλος μπορεί να λάβει το λόγο. Η ε, κυρία Μπότον, ευχαριστώ. Η Νορβηγία έχει ένα ηλεκτρονικό, μια ηλεκτρονική ενιαία θηρίδα όπου οι πάροχοι μπορεί να λάβουν πληροφορίες για το πώς μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στη Νορβηγία. Μιλάμε για, την, ε, για το PSC πρώτης γενεάς, το οποίο είναι διαθέσιμο έτσι ώστε να δώσει πληροφορίες σε παρόχους Τώρα, ποιοι παρέχουν αυτή την υπηρεσία, το όχτιν, ο φορέας που ασχολείται, έχει εντάξει αυτή τη διαδικασία στις, ε, στην άμεση εργασία της. Όλα αυτά έχουν περάσει στον Εθνικό Νόμο και η διαδικασία screening έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκλησή σας και γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα να σας μιλήσω για την εφαρμογή της ε, οδηγίας περιπηρεσιών στη Νορβηγία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ως προς το θέμα της ενιαίας θηρίδας του ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης είναι κάτι το οποίο έθιξε και η κυρία Γκέπχαρτ. σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμο στα νορβηγικά ή σε ποιες άλλες γλώσσες και σε ποιες άλλες γλώσσες. Και δεύτερο, ένα θέμα που θίγει από τις επιχειρήσεις, διότι έχετε και μια πολύ καλή έκθεση στο πακέτο σας που συνοψίζει το στάδιο μετάταξης ή μεταφοράς. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτά τα κέντρα ενίας εξυπηρέτησης σχετίζονται και με άλλους φορείς αδειοδότησης, δηλαδή μπορεί κάποιος να τελειώσει με, το, το με τα αιτήματά του μέσα ε, από αυτά τα κέντρα ενίας εξυπηρέτησης. Θα ήταν ε, ενδιαφέρον να το μάθουμε. Και αυτό ενδιαφέρει βεβαίως και άλλους συναδέλφους ως προς το πρώτο ερώτημα. Ξέρω ότι υπάρχει και σε άλλες γλώσσες, αλλά δεν ξέρω, ξέρω υπάρχει στα αγγλικά, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες γλώσσες. Και στα αγγλικά υπάρχει το, το σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης. Πώς θα εφαρμόσουμε ε, αυτή την οδεία και σε άλλες υπηρεσίες, δεν ξέρω σε πόσες υπηρεσίες θα ισχύσει, διότι εργαζόμαστε και με το Άλτη νέας γενιάς θα το βελτιώσουμε και θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η διασύνδεση του συστήματος. Επίσης έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα υπάρξει σύνδεσμος και εκεί. Ο κύριος Νέσφε. Ο κύριος Λεκρού θα ήθελε να παρέμβει σε... Ο κύριος Λεκού θέλει να παρέμβει σε αυτό το σημείο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ ναι, για να απαντήσω στο ερώτημα που θέσατε και να διευκρινίσω κάπως καλύτερα τη λειτουργία στη Γαλλία. Στη Γαλλία το Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο μέσω της νομοθεσίας ε, για τη μεταφορά της ε, οδηγίας ε, στο εθνικό δίκαιο, αλλά υπάρχει και ο ρυθμιστικός τομέας, ε, στον οποίο βέβαια αρμοδιότητα έχει κυρίως η κυβέρνηση. Έχει λοιπόν, είναι μια δουλειά μεγάλης κλίμακας, έχουν ήδη γίνει αρκετά πράγματα και υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα εντός της κυβέρνησης η οποία προσπαθεί να αξιολογήσει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προϋποθέτει η επιτυχής εφαρμογή της οδηγίας. Και όπως σας είπα είναι περίπλοκο γιατί είναι πολύ ευρύ το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εκτός από την πρωτοβουλία την, ε, των βουλευτών ε, δεν υπάρχει πρωτοβουλία των ε, τοπικών και περιφερειακών αργών. και θα ήθελα να ακούσω και από τους υπόλοιπους συναδέλφους και ειδικότερα από τη Γερμανία μήπως, δεν, μήπως υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίε σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατηδίων για παράδειγμα. Όσον αφορά τώρα την ενιαία θηρίδα, την ενιαία ε, εξυπηρέτηση, κάθε φορά που ένα, ηθικό, κάθε φορά που ένα ε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ε, θέλει να καταχωρήσει μία επιχείρηση, υπάρχει μία διπλή διάκριση μεταξύ μίας διοικητικής διαδικασίας η οποία θα είναι απλοποιημένη, πληροφορίες πολύ περισσότερες ε, συνεπώς ε, χάρη στο σύστημα αυτό και θα δώσει και τη δυνατότητα μάλιστα και στις άλλες χώρες, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να δουν ε, πώς μπορεί να γίνει η εφαρμογή της νομοθεσία στη Γαλλία. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστημα αποτελεσματικό το οποίο σιγά σιγά άρχισε να γίνεται συνήθεια στους Γάλλους, για να το πω έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τούν από την ε, Επιτροπή ε, Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Άλλο. Τελείως διαφορετικό θέμα και λίγο τεχνικό. Πολύ ενδιαφέρον ε, έχουμε τους βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ. Αναφέρατε, αναφέρατε και μία τηλεδιάσκεψη που έγινε και είπατε ότι αν το κοινοβούλια έχουν την, τον εξοπλισμό μπορούμε να το ξανακάνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε όσο πιο συχνά γίνεται. Ακόμη και αν τα κοινοβούλια δεν έχουν τον εξοπλισμό, στην ε, πρωτεύουσα υπάρχει ε, εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σίγουρα, και εκεί υπάρχει ο, ο απαραίτητο εξοπλισμό που να διευκολύνει την επικοινωνία. Θα πρέπει να επικοινωνούμε πολύ πιο συχνά και να έχουμε τέτοιου είδου ανταλλαγέ απόψεων. Εγώ θα, το, θα σας πρότεινα να το κάνουμε πιο συχνά Ακόμη και αν μπορείτε βέβαια δηλαδή και εσείς να είσαστε παρόντες εδώ συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που το θυμίζετε κυρία Τούν. Μπορεί να χρειαστεί να τον ενεργοποιήσουμε. Η κυρία Βερνιό. Μάλιστα. Ήθελα να πάρω το λόγο και επειδή πήρε το λόγο και ο Γάλλος συνάδελφος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε ε, παρόν και εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Πρόκειται για μια οδηγία πολύ περίπλοκη, όλοι το ανέφεραν και γι' αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό να συζητήσουμε. Είναι γεγονός ότι μου ε, μου πήρατε τα λόγια πραγματικά από το στόμα. Είναι γεγονός ότι από τη μία γίνονται πολλά πράγματα για την εφαρμογή της νομοθεσίας και από την άλλη υπάρχει έτσι μία λίγο αόριστη κατάσταση. Αναφερθήκατε κι εσείς ε, στους νόμους εξυγχρονισμού ε, της, ε, του τουριστικού κλάδου, της οικονομίας, των νοσοκομείων και μιλήσατε για τη σχέση αυτών με την οδηγία των υπηρεσιών και μιλήσατε και για τα νοσοκομεία ιδιαίτερος, κάτι το οποίο βέβαια δεν μου φαίνεται είναι του ιδίου επίπεδου με την οδηγία υπηρεσιών, ε, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με άλλου είδους πολιτικές. Βλέπουμε λοιπόν την σημασία και το περίπλοκο του πεδίου εφαρμογής. Ε, υπάρχουν και άλλα ε, και άλλες ιδιαιτερότητες, όλες αυτές οι φαιές ζώνες για τις οποίες μίλησε προηγουμένως και η κυρία Γκέπχαρτ επειδή έχουν κάποιες υπηρεσίες κοινή ωφελία εξαιρεθεί έχουμε κάνει κάποιους καταλόγους υπάρχουν κάποιες φαιές ζώνες ε, ε, για τις υπηρεσίες, ε, τις κοινωνικές, τις ιατρικές υπηρεσίες που πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν για την καθημερινή ζωή των πολιτών και για αυτά τα σημεία θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις και δυσκολίες εφαρμογής επιτόπου. Γι' αυτό θα χρειαστεί ακόμη περισσότερο να συζητήσουμε με όλους τους φορείς, ε, με τους ε, ε, εθνικούς βουλευτές, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ πολύ. And, uh, Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σεύτσικ. Όπως είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, 15 κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης ε, υπάρχουν ε, στην Τσεχία, 13 ε, στις διάφορες περιφέρειες και 2 στην Πράγα. Επίσης έχουμε και έναν ιστότοπο www.businessinfo.cz ε, ε, και μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας αυτής. Όσον αφορά την αξιολόγηση και την ευθύνη για την εφαρμογή της, ε, της οδηγίας αυτής, ο υπεύθυνο Υπουργείο είναι ε, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου στην Τσεχία. Πρόεδρος, το www.businessinfo.cz ε, υποθέτω ότι υπάρχει και στα αγγλικά, όχι μόνο στα τσεχικά. Ναι, υπάρχει στα τσεχικά και εν μέρη, όχι, ολόκληρα, όχι ολόκληρο, ε, στην, στα αγγλικά. Νομίζω και στα γερμανικά υπάρχει. Uh, good. Now, Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο για το ζήτημα αυτό των κέντρων εξυπηρέτησης, γιατί μας φαίνεται ότι είναι σημαντικό. Έχω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα τους Βρετανούς συναδέλφους που ήρθαν σήμερα το πρωί και με ενημέρωσαν. Τα Βρετανικά Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης άρχισαν ε, να λειτουργούν από το Δεκέμβριο 2009 και από το Φεβρουάριο και μετά λαμβάνουν αιτήματα για ενημέρωση, αιτήματα χίλια ε, το μήνα, 1300 ε, με τη μορφή τηλεφόρτωσης ε, των ηλεκτρονικών εντύπων. Μιλάμε για τεράστια νούμερα δεν ξέρω κατά πόσο ε, έχετε κι εσείς τέτοιου είδους αριθμητικά στοιχεία, αλλά θα θέλαμε να γνωρίζουμε και τέτοιου είδους δεδομένα, αν τα έχετε στη διάθεσή σας βεβαίως. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο για το συγκεκριμένο αυτό το θέμα, γιατί ξέρω και η κυρία Γκέπχαρτ θέλει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις αν δεν θέλει κανεί άλλο να πάρει το λόγο, να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ. Αλλά όπω σα είπα, τέτοιου είδου στοιχεία θα θέλαμε να τα γνωρίζουμε. Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση στον συνάδελφο από τη Γαλλία. Τι έγινε στην ε, Γερμανία και πώ ε, λειτουργήσε το ομοσπονδιακό σύστημα. Όντω, αυτό αποτελεί ούτως ή άλλως ε, δυσκολία για τη Γερμανία για τη δημιουργία των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης είναι αρμόδια τα κρατήδια από μόνα τους, αυτοτελώς αρμόδια. Ε, το Βερολίνο προσπάθησε να κάνει έτσι ένα συντονισμό, αλλά κατέρευσε, οπότε κάθε κρατήδιο τώρα έχει βρει μια δική του λύση για, τις, ε, για τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Ε, είναι κρίμα η αλήθεια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για τους ε, παρόχους υπηρεσιών από άλλες χώρες να βρούνε πού πρέπει να αποταθούν κτλ. Η ιδέα υπάρχει να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα, Απλώ πρέπει να βρούμε και τους κατάλληλου ανθρώπους. Στο δικό μου το, κρατήριο, το κρατήριο τη Βάδη Βιτεμβέργη, οι δύο εταίρειε στην συναυσπισμό δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για το σύστημα και υπάρχει διπλό σύστημα τώρα. Υπάρχει το σύστημα του κρατηδίου και υπάρχει και το σύστημα το περιφερειακό, της τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή. Και αυτό βέβαια είναι πρόβλημα. Αλλά δυστυχώ δεν μπορούσε να λυθεί αλλιώ. Στη Γερμανία λοιπόν όντω υπάρχει ανάγκη να λυθεί το θέμα αυτό έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν πρόσβαση στη γερμανική αγορά. Πρέπει να υπάρξει και ένα, μια κοινή πύλη, ένα πόρταλ, ώστε να μπορεί κανείς να ξέρει πού αποτείνεται όταν έχει κάποιο θέμα Καλό θα ήταν βέβαια να αρχίσει να λειτουργεί αυτό. Η κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει, γιατί δεν είναι αυτό που είχαμε φανταστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Και να σας θυμίσω επίσης ότι στην αρχική μου πρόταση της έκθεσης μου για την οδηγία για τις υπηρεσίες είχα προτείνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να... Μίλα λίγο φυσικά, σε παρακαλώ. Είχα προτείνει λοιπόν να, γίνει μια, να υπάρξει μια συντονιστική αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσει όλο αυτό να συντονιστεί. Βέβαια δεν ε, συμφώνησαν πολύ μαζί μου. Σήμερα έχω την εντύπωση ότι κρίμα που δεν τα καταφέραμε να έχουμε αυτή τη συντονιστική αρχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποφεληθούμε ίσως από τις βέλτιστες πρακτικές Ίσως ε, οι σημερινές ε, η σημερινή συζήτηση να είναι χρήσιμη, ελπίζω τουλάχιστον για το μέλλον. Ένα ερώτημα που έθεσε και ένα συνάδελφος. Υπάρχουν ήδη αριθμητικά στοιχεία. Πόσοι έχουν ε, στραφεί στην, ε, στα κέντρα νέα εξυπηρέτηση και σε ποιε γλώσσε έχει γίνει η ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, για τη δική μου τη χώρα είναι κρίμα γιατί συνήθως ε, τα περισσότερα ε, κέντρα εξυπηρέτησης βρίσκονται, είναι στα γερμανικά. Οπότε δεν έχει κανένας ε, το, δικαι... το... τη δυνατότητα, αν δεν μιλάει γερμανικά, να έχει πρόσβαση στην αγορά και τώρα προσπαθούμε να γίνει δίγλωσσο το σύστημα, να έχει και αγγλικά. Θα ήθελα να μου πούνε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τι γίνεται στα δικά τους, ε, στη δική τους επικράτεια. I'm sorry, interrupting you, but... Ε, λυπάμαι που σε διακόπτω, Εύελιν, αλλά έλεγα στη γραμματή ότι θα ήθελα η κυρία Μάρτιν Πράτ να μας πει ορισμένα λόγια. Είναι υπεύθυνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών και ίσως θα ήθελα να σχολιάσει ορισμένα από τα σημεία που εθίγησαν και να μας δώσει και ορισμένα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως προς το θέμα που συζητάτε επί του παρόντος, Δηλαδή η σύσταση ενιαίων κέντρων εξυπηρέτηση από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πω και δεν το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε ενώπιον εκπροσώπων από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να πω ότι έχει αναλυφθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα κράτη-μέλη και έχει επιτελεστεί πρόοδος. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα και δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε το γεγονός ότι από σήμερα υπάρχουν 22 λειτουργικά ε, σημεία ενίας εξυπηρέτησης και τα 5 που υπολείπονται ελπίζουμε να συσταθούν. Μιλάμε για ε, πρώτης γενεάς ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης που θα πρέπει να βελτιωθούν ανά το χρόνο. Μην ξεχνάμε όμως ότι μιλάμε για τα ε, σημεία τα οποία θα εκπροσωπούν ε, τις κυβερνήσεις, ε, της χώρες, θα παραμείνουν για δεκαετίες. Και αυτό αυτό είναι εξαιρετικό ως προς την εφαρμογή της οδηγίας. Γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη έχουν οργανώσει ευκαιρίες για να ανταλλάξουν απόψεις ως προς τη θέση εφαρμογή αυτών των ενιαίων σημείων. Δηλαδή, όρισαν ένα κοινό λογότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσπαθούν να ε, δώσουν στοιχεία και σε άλλες γλώσσες, όχι μόνο στην εθνική γλώσσα, αν και δεν προαπαιτείται από την οδηγία. Θα πρέπει λοιπόν να επενέσουμε τα κράτη-μέλη για αυτή την προσπάθεια. Πρόκειται για ένα μακρόπνοο σχέδιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι που έγινε, έληξε προθεσμία και πέρασε. Θα πρέπει να γίνεται μια συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και αυτό υπέρ των ΜΜΕ κυρίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενθαρρυντικά αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις όμως. Θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας σε σχέση με την διαδικασία screening, εξέτασης της νομοθεσίας ε, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό. Και επίσης να μας πείτε και την άποψή σας ε, για τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης συγκεκριμένα και για το λογότυπο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως νομικός πρέπει να σας πω ότι δεν βγαίνουμε να λέμε ε, για το λογότυπο, για το κατατεθέν σήμα, γιατί μόλις τώρα το ολοκληρώνουμε. Ε, θα είναι έτοιμο, πολύ σύντομα, Ελπίζουμε ότι θα προστατεύεται σύντομα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα σταματήσω εδώ, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Και το λογότυπο τα περισσότερα κράτη-μέλη το γνωρίζουν ήδη. Όσον αφορά τώρα την εξέταση της νομοθεσίας, ήταν ε, προϋπόθεση για την εφαρμογή της, της οδηγίας, γιατί όπως ήδη υπόθηκε, εκτός από την έγκριση οριζόντιας νομοθεσίας ε, για τις γενικές αρχές, ε, τα κράτη-μέλη έπρεπε να εντοπίσουν τις προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας που έπρεπε να προσαρμοστούν στην οδηγία. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια και έχει προσδώσει κάποιο βαθμό διαφάνειας που επίσης είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το καινούριο στο πλαίσιο της ε, οδηγίας ε, για τις υπηρεσίες. Ε, με μάτια εσωτερικής αγοράς είδαν τα κράτη-μέλη την ίδια τους την νομοθεσία. Στα κράτη-μέλη βέβαια που έχει ολοκληρωθεί η εξέταση. Για τα κράτη-μέλη που δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέτηση, δυστυχώς Κρίμα, αυτό είναι το μόνο που έχω να πω, γιατί ήταν προϋπόθεση για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην νομοθεσία. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σας. Αν θέλετε, ευχαρίστω να σας δώσω και άλλες πληροφορίες. Okay. Well, thank you very much Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Ναι, βεβαίως και μπορεί να υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις ε, από τους συναδέλφους. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Φαμπ ήθελε επίσης να κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Πράττα από την Κομισιόν για τη διαδικασία ελέγχου, θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα στους βουλευτές από τα κράτη-μέλη. Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν ασχοληθεί με το θέμα μέσω του screening για τις εθνικές δηλαδή διατάξεις οι οποίες μπορεί να μην είναι συμβατές με, τις, με την οδηγία. Ξέρουν οι πολιτικοί που έχουν εμπλακεί στην όλη αυτή τη διαδικασία ότι κάποιες, σε κάποιο επίπεδο κάποιες διατάξεις πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να προσαρμοστούν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο έπρεπε να είχα καλωσορίσει την κυρία Μάρτιν Πράτ νωρίτερα. Ζητώ συγγνώμη. Υπάρχουν και άλλοι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών που παρακολουθούν την κατάσταση. Αν θέλουν και εκείνοι να πάρουν το λόγο για το θέμα αυτό ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα της οδηγίας, ε, ευχαρίστως να τους ακούσουμε. Υπάρχει κανείς άλλος? Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Επειδή τα ενία αυτά κέντρα από το τέλος του 2009 θα πρέπει να εμπεριέχουν όλα τα σημαντικά στοιχεία καθώς και στοιχεία περί διοικητικής ε, ε, διεκπαιρέωσης. Ε, άκουσα και την άποψη των άλλων συνοδέλφων και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε δύο γλώσσες εκτός από τη γλώσσα της χώρας προέλευσης για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις, τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη χώρα η οποία θα ανοίξει τις πόρτες της στους ενδιαφερόμενους. Uh, yes, uh, thank you very much indeed for that. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, να ρωτήσει κάτι από τη Σουηδία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς, από σουηδικής πλευράς, είπαμε ότι θα έπρεπε να ληφθεί μια, απόσταση, μια απόφαση από το Κοινοβούλιο. Αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται πάντοτε σε επίπεδο ε, υπαλλήλων και είναι πολύ δύσκολο να εμπλέξουμε το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτήν την κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε εμείς να σας βοηθήσουμε σε αυτό, αλλά ενδιαφέρον είναι αυτό που μας είπατε. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο στο μέλλον ε, να το λάβουμε υπόψη, ώστε να συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια νωρίτερα στη διαδικασία στο μέλλον. Γιατί ήδη κάναμε μία συνεδρίαση σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες και έχουμε σκοπό να το κάνουμε πιο συχνά στο μέλλον. Oui, pour ne pas abuser, Ο κύριος Λεκού. Να μην ε, καταχραστώ τους, ε, της καλοσύνης σας και του χρόνου σας, απλώς... Ε, να απαντήσω στην ε, συνάδελφο ε, που με ρώτησε για τα νοσοκομεία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η νομοθεσία εφαρμόστηκε ακριβώς ε, βλέποντας πόσο ευρύ είναι το πεδίο της συγκεκριμένης οδηγίας. Γι' αυτό το έδωσα το, παρά, το, το παράδειγμα αυτό. Ε, συγγνώμη για αυτή τη γαλλογαλλική παρατήρηση, απλώς προσπάθησα να σας δείξω το περίπλοκο της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πριν πάρει το λόγο και πάλι η κυρία Γκέπχαρτ, μήπως θέλει κανείς άλλος να ρωτήσει τίποτα. Μιλήσαμε και για την απλοποίηση των ε, εσωτερικών κανόνων. Δεν ξέρω αν θεωρήσατε ότι όλη η όλη διαδικασία βοήθησε την απλοποίηση της διαδικασίας, της διαδικασίας σας. Δεν έλαβα απάντηση σε αυτό. Ξέρω κυρία Γκέπχαρντ ότι παρακολουθήσατε πολύ το ζήτημα αυτό. Μήπως θέλετε να αναφερθείτε πιο πολύ σε αυτό το θέμα ή σε οτιδήποτε άλλο. Για τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Είναι όντως από τα πιο σημαντικά στο, στις, για την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες, γιατί πραγματικά προωθεί και διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές. Είναι διοικητικό θέμα όμως αυτό, που μάλλον δεν πολύ συζητείται και στα κοινοβούλια, το οποίο όμως παρόλα αυτά είναι σημαντικό. Και για διάφορους λόγους είναι σημαντικό αυτά τα κέντρα να τα μελετήσουμε ενδελεχώς. Καταρχήν γιατί είναι τα κέντρα που έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται οι πάροχοι υπηρεσιών για να σέβονται τους κανόνες που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Να του δώσουν δηλαδή τι πληροφορίε, να μην του αφήνουν μόνο του να ψάχνουν, μόνο να ψάχνουν πώ είναι το εργατικό δίκαιο στην τάδε χώρα, τι πρέπει να κάνω για την περιβαλλοντική προστασία κτλ. κτλ. Όλοι λοιπόν αυτοί οι κανόνε που ισχύουν στα κράτη-μέλη ε, εξακολουθούν να υφίστανται και να ισχύουν και θα πρέπει να συμβαίνει αυτό εφόσον το επιθυμούν τα κράτη-μέλη. Δεν, χρειάζεται δηλαδή να τα διαγράψουμε όλα επειδή ξαφνικά υπήρξε η οδηγία για τι υπηρεσίε. Αυτό είναι λοιπόν το ένα για τις πληροφορίες. Το δεύτερο. Απλοποιείται πάρα πολύ η, διοικητική, η πρόσβαση στις διοικητικές αρχές. Εγώ μπόρεσα στη Γερμανία να συζητήσω με αρκετούς που μου είπαν ότι για μας ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν είδαμε ότι μέσω όλου αυτού του κοινού συντονισμού καταφέραμε να εξυγχρονίσουμε και τη δική μας τη, διοίκηση, γιατί είδαμε πόσο δύσκολο είναι να έχουν η πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες οι επιχειρήσεις, οπότε, και δεν μιλούμε μόνο για, τους, ε, για ε, εκτός Γερμανίας παρόχους υπηρεσιών, αλλά και για τους Γερμανούς. Και θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο και για άλλους τομείς. που πρέπει να εφαρμοστούν μέσω τη οδηγία για τι υπηρεσίε, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση. Αυτό είναι το, το δεύτερο, γιατί αυτά τα κέντρα ενιαία εξυπηρέτηση είναι τόσο σημαντικά. Και τρίτον, απλούστευση για του παρόχου υπηρεσιών. Αυτό είναι σαφέ, θεμητό και βεβαίω υπάρχει και το θέμα των γλωσσών με τι οποίε μπορεί να έχει κανεί πρόσβαση στην αγορά και χαίρομαι που η Κομισιόν έχει βγάλει αυτό το λογότυπο, το κοινό, το... για να υπάρχει έτσι μια γενική διαφάνεια. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο ακόμη συζητείται, θα μπορούσε να συζητείτε στα κράτη-μέλη, οι πληροφορίες Προ του παρόχου. Δηλαδή να έχουν έναν ε, συνομιλητή ο οποίο θα είναι το κέντρο ενιαία εξυπηρέτηση και εγώ σε πολλέ συζητήσει που έκανα με επιχειρήσει, διαπίστωσα ότι πολλέ μικρομεσαίες επιχειρήσει δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα κέντρα εξυπηρέτηση, δεν χρησιμοποιούν λοιπόν αυτέ τι δυνατότητε, αυτέ τι ευκαιρίε. και γι' αυτό ακριβώ είναι το πιο, γι' αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικά τα κέντρα αυτά. Και στρέφομαι προ την Κομισιόν θα μπορούσατε ίσως να κάνετε μια ενημερωτική εξτρατεία από κοινού με τα κρατημέλη, έτσι ώστε να το γνωρίζουν καταρχήν οι επιχειρήσεις, ποιες δυνατότητες υπάρχουν, ποιες ευκαιρίες υπάρχουν στον τομέα αυτό για την πρόσβαση στην αγορά και πού κανείς μπορεί να στραφεί όταν χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες. Να μπορέσει δηλαδή αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί, να μην είναι μόνο θεωρητικό. Αυτά έτσι, για να σας διευκρινίσω λίγο τα πράγματα. Και γι' αυτό χρειάζομαι και τη βοήθεια ε, των, συναδέλφων από τα Εθνικά Κοινοβούλια, έτσι ώστε αυτό το εργαλείο που δημιουργήθηκε να χρησιμοποιηθεί και να μπορέσει επιτόπου να διευκολύνει, να φέρει κάτι θετικό στην, καθημερινή, ε, στην καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών. Δεν, κάνουμε, ε, δεν εκπονούμε πολιτική μόνο για του σκοπού τη πολιτική. θέλουμε να προσφέρουμε στου Ευρωπαίου πολίτε και θέλουμε να φροντίσουμε ότι για, τις, για την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών θα, τηρου, θα τηρηθούν όλοι αυτοί οι κανόνες και θα απλοποιηθούν τα πράγματα. Να μπορέσουμε δηλαδή να σπάσουμε και μονοπόλια κτλ. Αυτά λοιπόν κάποια σημεία για τα κέντρα ενίας εξυπηρέτησης. Αν δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να θέλει το λόγο, για αυτά τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης. Ίσως να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Θα έκανα μια πρόταση. Ήρθαμε σε επαφή με το γραφείο του κυρίου Μπαρνιέ να δούμε αν μπορεί να έρθει λίγο πιο νωρί. Ακούστηκαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα σημεία και ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα και να τα πούμε λίγο ατύπως, γιατί και η κυρία Μάρτιν Πράτ και άλλα μέλη τη Κομισιόν είναι εδώ και εσεί είστε εδώ, οπότε ίσως να κάνουμε ένα ε, διαλυματάκι μέχρι τις 5 και 4. Ο Επίτροπος θα έρθει 5.30-6 παρά 20 για να κάνουμε τις επίσημες συζητήσεις και να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Και βεβαίως και εσείς ίσως να θέλετε να μας θέσετε κάποια θέματα. Και θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να μπορούμε να τα διαχειριστούμε όταν θα έρθει και ο επίτροπο. Θα ζητήσουμε και τη βοήθεια της κυρίας Μάρτιν Πράτ. Και επειδή είσαστε και λίγο μακριά, έχετε κάτσει εκεί λίγο πίσω, ε, να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Οπότε, ε, αν συμφωνείτε, κάνουμε ένα διαλυματάκι και τα ξαναλέμε στις 5 και 4. Να τεντώστε και λιγάκι τα πόδια σας, να ξεκουραστείτε. Και μετά, στον τελευταίο γύρο συζητήσεων, θα δώσουμε το ρόλο στην κυρία Γκέπχαρτ για να κάνει μια εισαγωγή. Θα ακούσουμε κάποια ε, καταληκτικά σχόλια που θέλετε, αν θέλετε να κάνετε. Εντάξει, Εύελιν. Ωραία. Οπότε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νερά ή ποτά έξω. Ας μεταφερθούμε όλοι προς τα έξω για να τα πούμε και στις 5 και 4 ξαναρχόμαστε στην αίθουσα. Uh, so, ladies and gentlemen, I think um, I suggest uh, and um, Να συνεχίσουμε. Και να δούμε μήπως υπάρχει τίποτε άλλο που προέκυψε κατά τη διάρκεια του διαλύματος και εγώ είχα τη δυνατότητα να συστηθώ σε πολλούς ε, από τους συναδέλφους. Και όπως ξέρετε, έχουμε διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου που ασχολούνται με επιμέρους θέματα που άπτονται και του δικού μας και θα ήθελα να ξαναδούμε το, την εμβέλεια της οδηγίας και ίσως η Εύελιν Γκέπχαρτ θα μπορούσε να μας πει ορισμένα ε, λόγια. Θα θέλαμε να μας πείτε κατά πόσο βρίσκεται χρήσιμες αυτές τις συνεδριάσεις και αν υπάρχουν άλλα θέματα που ενδεχομένως σας απασχολούν σε σχέση, που, σε σχέση με θέματα που καλύπτουμε εμείς ως προς την εσωτερική αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα εργασίας για την Κομισιόν, για την, ε, συγγνώμη, για την Επιτροπή μας για τους επόμενους 20 μήνες και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχουν άλλοι τομείς που σας ε, απασχολούν. Θα ήθελα να ε, μας πείτε αν υπάρχουν τέτοια θέματα. Ο κύριος Μπαρνιέ είναι κάθοδον και θα μας μιλήσει για επιμέρους θέματα που άπτονται τις οδηγίες. Η κυρία Πράτ είναι εδώ, η κυρία Μαρτίν Πράτ από την Κομισιόν είναι εδώ και ίσως θα ήταν σκόπιμο να δώσω το λόγο για ορισμένα συμπερασματικά σχόλια. Η Εύελιν θα ήθελε κάτι να μας πει ε, εν είδη εισαγωγής. και θα ήθελα να μου πείτε όποιος επιθυμεί το λόγο να μου το κοινοποιήσει. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω, τα οποία μου αναφέρθηκαν στο διάλειμμα και τα οποία έχουν σχέση και με το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμογή του πεδίου εφαρμογής. Το ένα είναι ένα σημείο για το άρθρο 1, παράγραφος 6 όπου λέει ότι αυτή η οδηγία δεν άπτεται του εργατικού δικαίου. Δηλαδή, οι διατάξεις ε, για, για τις ε, συνθήκες ε, απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων και των υγειονομικών και των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και εργοδοτών τα οποία, οι οποίες ορίζονται από το κράτος μέλος, δυνάμει του ε, εθνικού του δικαίου, μπορούν να εφαρμόζονται. Και επίσης η οδηγία αυτή δεν άπτεται των διατάξεων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτή η διάταξη νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Γιατί υπήρξε έτσι αρκετά μεγάλος φόβος στα κράτη-μέλη για το ότι αυτό το αυτή η νέα οδηγία θα, θα, θα έκανε τις διατάξεις των κρατών μελών παροχημένες. Αυτό δεν συμβαίνει βέβαια. Έγιναν μεγάλες συζητήσεις μακροσκελής για το αν μπορούμε να το συμπεριλάβουμε ή όχι αυτό. Το συμπεριλάβαμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι εδώ δεν μιλούμε για το ότι θα υπάρξει πρόβλημα ή θα τροποποιηθεί το εργατικό δίκαιο του κράτους μέλους. Ούτως ή άλλως αυτό το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Ξέρω ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά ίσως ε, να μπορέσει έτσι να διαλευκανθεί γιατί η συμπαιγνία μεταξύ της, υπηρεσίας, της οδηγίας για, την υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες και όλες, τις, και όλες οι υπόλοιπε οδηγίες φυσικά έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν. Και πολύ σημαντικό επίσης είναι το πεδίο εφαρμογής. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά είχε προτείνει αυτές οι υπηρεσίες και η οδηγία για τις υπηρεσίες να <clears throat> ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των καθαρά εμπορικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή οδηγία και των υπηρεσιών κοινού ε, οικονομικού συμφέροντος που χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Για παράδειγμα, οπτικοακουστικά, υπηρεσίες μεταφορών, κοινωνικές υπηρεσίες, άλλες δραστηριότητε δραστηριότητες συμβολεογράφων, ε, κλητήρων κλπ. Ε, κάποια παραδείγματα για του άρθρου 2 σας αναφέρω. Αυτά εξαιρέθηκαν. Και επίση εξαιρέσαμε τα τυχερά παιχνίδια, γιατί είπαμε ότι δεν είναι υπηρεσίε κοινωνικού χαρακτήρα, ούτε κοινού κοινωνικής, ε, κοινωνικών υπηρεσιών αλλά ειδικέ υπηρεσίες. Ούτε δηλαδή στις γενικές υπηρεσίες μπορούν να εμπέσουν. Προστασία λοιπόν, εδώ περιλαμβάνεται και η προστασία για, από το οργανωμένο έγκλημα. Και εν μεταξύ και το δικαστήριο είπε σαφώς ότι είχατε, είχατε που το, που το διαχειριστήκατε έτσι το θέμα γιατί έπρεπε να δημιουργηθούν κάποιες ειδικέ διατάξεις για τα κράτη-μέλη. Μία από τις βασικές συζητήσεις και τα αμφιλεγόμενα σημεία που υπήρξαν στο ιστορικό του Κοινοβουλίου και στα κράτη-μέλη ήταν ο υποκλεισμό των ε, υπηρεσιών κοινού οικονομικού συμφέροντος, πώς μπορούν αυτές να αποκλειστούν και με βάση ποια κριτήρια. Στη συμβαστική πρόταση, στην οποία καταλήξαμε, βεβαίως υπάρχουν και αδύναμα σημεία, το παραδέχομαι ε, και οι συμβασμοί πάντα είναι συμβασμοί. Το θέμα είναι πώς θα ερμηνευθούν από τα κράτη-μέλη και πώς θα τα διαχειριστούν τα κράτη-μέλη. Και θα με ενδιαφέρει πολύ να δω πού υπάρχουν προβλήματα. Πού έχετε μείνει πίσω σε σχέση με τα δύο αυτά σημεία που σας ανέφερα. Δηλαδή, καταρχήν σεβασμός του εργατικού δικαίου και αποκλεισμός των υπηρεσιών κοινού οικονομικού συμφέροντος. Νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει και ένα εγχειρίδιο Διάβασα εγώ κάποια πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ και ιδιαίτερα. Γιατί είπα δύο λεπτά. Το κοινοβούλιο αποφάσισε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, σε έναν τομέα, στην υγεία ας πούμε, στα νοσοκομεία, τα οποία ξερούνται, οι υπηρεσίες υγείας ξερούνται. Στο νοσοκομείο λοιπόν παρέχονται και κάποιες υπηρεσίες όπως εστιατόρια, καντίνες, φαγητό για τους ε, ασθενείς. Και αυτοί πρέπει να φάνε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβάζει από την δική μας ε, πρόταση ότι, ερμηνεύει μάλλον από τη δική μας πρόταση, ότι αυτό δεν ανήκει στις υπηρεσίες υγείας, αλλά θεωρείται εμπορική δραστηριότητα. Ειλικρινά έμεινα με το στόμα ανοιχτό με την ερμηνεία που έδωσε η Κομισιόν. Γιατί αυτές οι υπηρεσίες της σύντησης των ε, ασθενών που είναι πολύ ειδικέ οι συνθήκε, οι διατροφικέ συνήθειε, οι δίαιτε που πρέπει να ακολουθήσουν κτλ. Ανάλογα με την ασθένεια που έχει ο καθένα. Όλο αυτό είναι κομμάτι του συστήματο υγεία. Δεν είναι κομμάτι του εμπορικού, των εμπορικών υπηρεσιών. Ε, Αυτέ είναι κάποιε έτσι συνέπειε που τελικά παίζουν ρόλο. Και θα με ενδιαφέρε να μου πείτε, στα κράτη-μέλη η συζήτηση αυτή προ τα πού κινήθηκε. Έγινε καταρχήν. Πώς το ερμηνεύσατε εσείς και ποια είναι τα προβλήματα και αν λύθηκαν τα προβλήματα αυτά. Μιλούμε δηλαδή για αυτά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και πώς μπορούμε μέσα από ένα κείμενο, να, ακόμη και συμβαστικό, να διαβάσει τελικά ό,τι θεωρεί ότι πρέπει να διαβάσει. Πραγματικά εγώ δεν το είχα σκεφτεί ότι μπορούσε να ερμηνευτεί έτσι η πρότασή μας όταν το είχαμε συζητήσει και με, από συζητήσεις με τους συναδέλφους στο κοινοβούλιο και από άλλες ομάδες, είδα ότι είχαν και αυτοί αντίστοιχη αντίδραση με μένα. Οι κοινωνικές, α, οι κοινωνικές υπηρεσίες εξαιρέθηκαν και τώρα γιατί μιλούμε ας πούμε για τα μικρά παιδιά. Μάλλον εντάξει, δεν είμαστε και όλοι τη ίδια αποψή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Και περιμένω να δω τι θα πούνε και οι συνάδελφοι. Okay, yes. Uh, Mrs. Mrs. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θυμηθήκατε το όνομά μου. Όταν πρόκειται για την αγορά εργασίας, σας το είπα και προηγουμένως ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν ήταν πια οδηγία Μπόλκενστάιν. Αλλά προσπαθήσαμε εμείς στη Σουηδία να αλλάξουμε την νομοθεσία, να προβλέψουμε κάποιες εξαιρέσεις ε, και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι Κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μας είπαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος για να ελέγξει ακριβώς ε, τι γίνεται με τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Και καταφέραμε να απομακρύνουμε κάποια στοιχεία της ε, νομοθεσίας που δεν ήταν πολύ ευνοϊκά και καταλήξαμε σε ορισμένα σημεία για τα οποία εκφράσαμε κάποιες ανησυχίες και το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να ασχολείται με το ζήτημα αυτό και ε, στο πλαίσιο της εξέτασης εφαρμογής οδηγίας. Ε, διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα. Ή θα έπρεπε να διευρευνήσουμε κάποιους, κάποιες άλλες διόδους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας στη Σουηδία να καταφέρουμε να κάνουμε μια συνεκτίμηση όλων αυτών των πραγμάτων με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με το δικό μας Κοινοβούλιο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πώς ακριβώς ε, θα συνεχίσουμε. Η ανταλλαγή απόψεων πάντως είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια που θέλει να πάρει το λόγο, γιατί ε, ο κύριος Φαμπ και η κυρία Ράπτη θέλουν να πάρουν το λόγο. Κύριε Φαμπ. Ευχαριστώ, Σπάνια διαφωνώ με την κυρία Γκέπχαρτ, αλλά τώρα θα το κάνω. Στο 2F, στο άρθρο 2F, γίνεται σαφής αναφορά σε υπηρεσίες ανεξάρτητα από το αν ε, ε, προσφέρονται α, σε, εντός των, ε, του συστήματος υγείας. Δηλαδή η καθαρίστρια ή η ομάδα η καθαριστριών ή το φαγητό που προσφέρεται στα νοσοκομεία, η σύντηση. Είναι μια υπηρεσία που δεν είναι ιδιαίτερη για τον τομέα της υγείας. Γι' αυτό θα συμφωνήσω με την... Ε, με την Κομισιόν που λέει ότι θα πρέπει να έχουν κάποιες, να έχουν κάποια συνάφεια με τον τομέα τη υγεία οι, προ, οι υπηρεσίες αυτές για να μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής. Εντάξει, τώρα ένα άνθρωπο που έχει μια ειδική, μια ασθένεια που πρέπει να φάει κάτι πολύ συγκεκριμένο, εντάξει, υπάρχουν και ειδικέ περιπτώσει. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να εμπίπτουν. Ελπίζω να με υποστηρίξουν και άλλοι. Ευχαριστώ. Ωραία. Ενδιαφέρουσα μένετε τη συζήτηση. Έχουμε και την οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες, που επίσης επηρεάζει κάπως τα πράγματα. Αλλά η παροχή υπηρεσιών κοινού οικονομικού συμφέροντος καλύπτεται από πιο ισχυρέ ασφαλιστικέ δικλείδε, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και σε σχέση με τις προμήθειες. Ο κύριος Μπαρνιέ έρχεται. Η κυρία Ράπτη, καλώς ορίσατε και πάλι να σας δώσουμε το λόγο και μετά θα ακούσουμε οποιονδήποτε άλλο θέλει από τα κοινοβούλια να παρέμβει πριν έρθει ο κύριος Μπαρνιέ. Κυρία Ράπτη. Υποθέσω κύριε Πρόεδρε ότι μπορώ να μιλάω μέχρι να έρθει ο κύριος Μπαρνιέ. Τόση ώρα. <laughs> ε, όχι απαραίτητα τόση ώρα σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος που έλειψα είχε σχέση και με την συνεδρίαση που γίνεται εδώ. Είχα πάει στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου είμαι κύριο μέλος, και που εκεί υπήρχε ακρόαση του κυρίου Άντορ. Ε, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχει άμεση σχέση της εσωτερικής αργοράς και των α, δικαιωμάτων και της προστασίας των εργαζομένων. Ε, έχω λοιπόν να σας πω τα εξής. Δεν θέλησα να ζητήσω και προηγουμένως το λόγο γιατί ακριβώς νόμιζω ότι έπρεπε να μιλήσουν οι εκπρόσωποι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το πρώτο που θέλω να πω και θέλω να το πω με υπερηφάνεια είναι ότι τώρα που εμείς συζητούμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο για την οδηγία αυτή για τις υπηρεσίες, στη χώρα μου, στην Ελλάδα, που ξέρετε τι συμβαίνει μην τα ξαναπώ, ψηφίζουμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο την, μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά κυρίως και για το Εθνικό Κοινοβούλιο και την Ελλάδα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Ωστόσο θα ήθελα να τονίσω δύο ακόμη πράγματα. Το ένα είναι ότι εφαρμόζοντας την οδηγία για τις υπηρεσίες θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας την προστασία των εργαζομένων και ταυτοχρόνως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, νομίζω, και την υπόθεση της αναλογικότητας. Άκουσα προηγουμένως με προσοχή και τον κύριο Σουάμ ε, σε σχέση με τη σύντηση. Αυτό που ε, σκέφτομαι είναι ότι ο τομέας της υγιεινής διατροφής έχει άμεση σχέση με την υγεία γενικώ, πολύ δε περισσότερο με την υγεία των ανθρώπων που αναγκάζονται να μπουν στα νοσοκομεία. Άρα, ερωτηματικό. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να έχει προσεκτικό διαιτολόγιο μόνο κάποιος ο οποίος μπαίνει σε ένα νοσοκομείο επειδή πάσχει από το στομάχι του, για παράδειγμα. Νομίζω ότι ίσως να έχει ανάγκη αυτός που μπαίνει και επειδή έχει κάνει μια εγχείρηση καρδιάς ή αυτός που έχει σπάσει ένα πόδι και άρα πρέπει να χάσει βάρος. Λέω, μερικές σκέψεις που έχω στο μυαλό μου ε, είναι λίγο περίεργες, βλέπω ότι κάνει κάποιες γκριμάτσες ο πρόεδρος, <laughs> αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα συζητάμε όλα για να μπορέσουμε να φτάνουμε στα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα. Ε, και κλείνω λέγοντας ότι πιστεύω πως έχουμε ανάγκη περισσότερο από όλους στο επίπεδο της εσωτερικής αγοράς αυτούς που την νομιμοποιούν. Και αυτοί που νομιμοποιούν την εσωτερική αγορά, το θέμα των υπηρεσιών και την καλή λειτουργία της δεν είναι άλλοι από τους πολίτες και τους καταναλωτές που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ναι, μπαίνουμε σε, κάποιες, σε κάποιους λεπτομερείς τομείς της συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων ε, για όλα τα ζητήματα που καλύπτει η οδηγία αυτή και νομίζω ότι είναι σαφές πλέον ότι είναι εξαιρετική ε, εξαιρετικά ευρύ θέμα και είναι κάτι που θα επηρεάσει όλους τους πολίτες σε μεγάλο βαθμό. Επίσης θα έχουμε και πολλές δυνατότητες, θα δώσουμε πολλές δυνατότητες στους πολίτες με διάφορους τρόπους ε, να εισακουστούν και εκείνοι. Είναι κάτι το οποίο δεν, δεν ε, το συζητήσαμε πολύ. Η προώθηση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, ε, η διαθεσιμότητα των πληροφοριών μέσω των κέντρων νέας εξυπηρέτησης είναι δυνατότητα, σημαίνουν δυνατότητα για τους πολίτες να ε, ιδρύουν επιχειρήσεις ε, και είναι κάτι το οποίο απευθύνεται κυρίως ε, στις μικρές επιχειρήσεις και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ευκαιρίες στη διάθεση των πολιτών πλέον. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μόνο ότι τις γνωρίζουν τις ευκαιρίες αυτές οι πολίτες. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε σε μία πρόταση για μία έκθεση του κυρίου Γκρέκ, μία έκθεση που επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, για ε, την εσωτερική αγορά, τους πολίτες και τους καταναλωτές είναι κάτι το οποίο ε, γίνεται παράλληλα ε, από τον καθηγητή κύριο Μόντι. Θα υπάρξει και μια η εισήγηση του κυρίου Μπαρνιέ και ενδεχομένω να θέλετε να τον ρωτήσετε σε σχέση με τη μελλοντική στρατηγική ολοκλήρωση ετορική αγορά, γιατί μα ενδιαφέρει πάρα πολύ όχι απλώ να είμαστε μια παθητική κοινοβουλευτική επιτροπή που περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη στείλει οδηγίε για να τι εξετάσει, να τι παρακολουθήσει. Θέλουμε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και την πολιτική ατζέντα. Και γι' αυτό θέλουμε τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και γι' αυτό ακριβώς ε, αυτό που προκύπτει από τη σημερινή μα συζήτηση είναι ότι η σημασία ε, συζήτησης ε, μαζί σας σε νωρίτερο στάδιο είναι πολύ σημαντική γιατί είναι μια πρόταση που αποφασίστηκε ήδη το 2006. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ο διάλογος μαζί σας. Πριν έρθει ο Επίτροπος Μπαρνιέ, μήπως θέλει κανείς να πάρει το λόγο από την Ορβηγία, ο συνάδελφος. Συγγνώμη, δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά σας, είστε πολύ μακριά. Κύριε Νέσφικ. Ευχαριστώ από νορβηγικής πλευράς ε, θα ήθελα απλώς με αυτή την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω διότι μας επιτρέψατε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συνεδρίαση. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι κοινέ συνεδριάσεις διότι έτσι έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε θέματα με βουλευτές από άλλες χώρες και ιδιαίτερα ε, από άλλα ε, κράτη, από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μία ευρύτατη συζήτηση και θα έχουμε και στο μέλλον έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα σοβαρά ζητήματα πριν από την τελική γνωμοδότηση. Πριν από την τελική σύνταξη δηλαδή παρόμοιων οδηγιών. Θα πρέπει να δούμε τις δυνατότητες που διανοίγονται από παρόμοιες οδηγίες και χωρίς να εστιάσουμε την προσοχή σε προβλήματα που μπορεί ειδικά να ανακύψουν στο μέλλον. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας επιτρέψατε να συμμετάσχουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα ίσως και αργότερα να λάβουμε το λόγο και σε μελλοντικές συνεδριάσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα σχόλια καταληκτικά προς στιγμή και ίσως έχουμε τη δυνατότητα για ορισμένες τελευταίες ερωτήσεις αργότερα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, Μισελ Μπαρνιέ, τον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα εσωτερικής αγοράς. Χαιρόμαστε που παρευρίσκεστε εδώ και θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το σημερινό μας θέμα και να δεχτείτε και ορισμένες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί ήρθατε λίγο νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο. Ξέρουμε ότι είσαστε χρονικά πιεσμένος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να μας πείτε τις δικές σας απόψεις για τη μεταφορά της οδηγίας περί υπηρεσιών και μηνύματα προς τα Εθνικά Κοινοβούλια που είναι παρόντα εδώ, καθώς και προς τα μέλη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω στο τέλος ε, της ε, κοινής αυτής συνεδρίασης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Χαίρομαι βέβαια για πολλούς λόγους, ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως ε, είναι στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και μάλιστα λίγο νωρίτερα όπως μας ζητήσατε και δεύτερον χαίρομαι πολύ γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτήν την αίθουσα. Είχα πολλές φορές τη δυνατότητα να έρθω γιατί ήμουν μέλος της Επιτροπής Και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, και από την ε, Γερουσία ε, των κρατών μελών ε, ότι ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ μάλιστα είχα αυτό το ρόλο στη χώρα μου πάνω από 20 χρόνια και πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς μια κοινή δουλειά, μια συνεργασία μεταξύ ευρωβουλευτών και εθνικών ε, ε, κοινοβουλίων. Γι' αυτό λοιπόν για τα επόμενα πέντε χρόνια έχω πάρα πολύ, έχω, έχω ε, σκοπό πολλές φορές ε, να ε, έρθω σε επαφή με τις αρμόδιες επιτροπές σε όλες τις πρωτεύουσες, το έκανα και το 2004 και θα το ξανακάνω κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Και έχω και ένα λόγο παραπάνω μάλιστα να το κάνω, γιατί τα θέματα ε, της αρμοδιότητός μου είναι ζητήματα όλα συναπόφασης. Ε, ο νομοθέτης, ο Ευρωπαίος και ο Εθνικός ε, έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίζει. Και όταν μιλάω για ουσιαστικό ρόλο των βουλευτών, θα ήθελα να πω ότι αναφέρομαι και στο ρόλο των Ευρωβουλευτών, ας πούμε, της κυρίας Γκέμπχαρτ στην έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες, που είναι και το αντικείμενο της σημερινής σας συνεδρίασης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον ε, πρόεδρο, τον κύριο Χάρμπουρ, για την σημερινή πρωτοβουλία και να σας πω ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια μπορείτε να στηριχθείτε σε μένα, θα είμαι διαθέσιμος πάντοτε για αυτόν τον διάλογο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί η οδηγία που είναι αντικείμενο της σημερινή συζήτηση είναι σημαντική. Κοιτάξτε, είναι τεράστιο το εγχείρημα της μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο πολλές φορές ε, το διαπιστώσαμε στην αρχή της ε, μακρόχρονης διαδικασίας βελτίωσης της οδηγίας. Βελτιώθηκε πολύ αυτή η οδηγία γιατί ήμουν μέλο και τη επιτροπή πρώτη που έκανε την πρόταση αυτή και όπως κάθε πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι βελτιώσιμη. Και βεβαίω βελτιώθηκε πάρα πολύ μέσω τη ε, κοινοβουλευτική ε, εργασία. Όμω, ε, επί τη ουσία, μιλάμε για ένα οικονομικό ζήτημα τεράστια σημασία και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι βάσει των υπολογισμών των υπηρεσιών μου, που επιβεβαιώθηκαν κιόλα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ωφέλη της σωστής εφαρμογής, της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας στα 27 κράτη-μέλη είναι μεταξύ 60 και 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, ε, μεταξύ 60 και 140 ε, δισεκατομμυρίων ε, ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για 1,5% επιπλέον ανάπτυξης. Και θα ήθελα να πω ε, στους εθνικούς βουλευτές που βρίσκονται εδώ ότι είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα που διακυβεύεται και πρέπει να εξεύρουμε νέους μοχλούς ανάπτυξης Όπω αυτό, Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδου μοχλή στο πλαίσιο τη οδηγία για τις υπηρεσίε, Και για ποιο λόγο είναι σημαντική αυτή η οδηγία. Δεν είναι μια οδηγία σαν τι υπόλοιπε όχι εντελώς τουλάχιστον. Είναι μια πρόκληση άνευ προηγουμένου για τα κράτη-μέλη, εκτός ε, από την ομοθετική εργασία ε, που χρειάζεται ε, για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Επιζητά επίσης την ενιαία θηρίδα, για παράδειγμα, για, τις, για την γραφειοκρατία, για τις διαδικασίες τις διοικητικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρχή ε, αφιέρωσε πολύ σημαντικούς πόρους ε, για να υποστηρίξει τεχνικά τα κράτη-μέλη. Και πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την εφαρμογή και τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Η προθεσμία ήταν 28 Δεκεμβρίου 2009 για τη μεταφορά, όπως γνωρίζετε. Τέσσερις μήνες μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, ε, μπορώ να ε, κάνω έναν απολογισμό ε, χωρίς ε, να παραλείψω βέβαια ότι διαπίστωσα την ε, καλή συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και Κρατών Μελών καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Υπάρχει κάποιο είδους αντίκτυπος εσωτερικής αγοράς λόγω του μοχλού που αποτελεί οδηγία για τις υπηρεσίες σε επίπεδο εθνικών διοικήσεων. Για παράδειγμα στη Σουηδία 3 και 4 Ιουνίου θα μεταβώ στη ε, Σουηδία στο πλαίσιο κάποιων ε, άλλων αρμοδιοτήτων μου. Θα αρχίσω 3-4 Ιουνίου τις επισκέψεις τις οποίες ε, σας είπα ότι θα κάνω σε όλες τις πρωτεύουσες για να συναντήσω τους αρμόδιους ε, υπουργούς, ε, ε, τους αρμόδιους για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής, όπως επίσης και την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα ή των δημοσίων προμηθειών. Είναι ζητήματα για τα οποία θέλω να επιβεβαιώσω, όχι μόνο με τους, σε συναντήσεις μου με τους υπουργούς, αλλά και με τους υπαλλήλους που έχουν αναλάβει, τους αξιωματούχους που έχουν αναλάβει την εφαρμογή τους. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας σωστός τρόπος ε, λειτουργίας και περιμένω ότι από αυτές τις ε, επισκέψεις ε, θα προκύψει ε, στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών ε, ε, αρχών μια καλύτερη κατανόηση της, της κατάστασης που απορρέει από τις εν λόγω οδηγίες. Τρία βασικά στοιχεία σε σχέση με την οδηγία. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την έγκριση και την τροποποίηση των ισχυουσών νομοθεσιών. Αυτή τη στιγμή 19 κράτη έχουν εγκρίνει την οριζόντια νομοθεσία μεταφοράς ε, στο εθνικό δίκαιο σε τέσσερα κράτη ε, αυτή τη στιγμή ε, βρίσκεται στο Κοινοβούλιο, ενώπιον του Κοινοβουλίου, του Εθνικού Κοινοβουλίου. Πέντε κράτη-μέλη και τα δύο ακόμη κράτη-μέλη που δεν έχουν ξεκινήσει ολοκληρώνουν αυτήν την σημαντική νομοθετική δουλειά και ελπίζω ότι κάθε ένας από εσά μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη δέσμευση των κρατών μελών ε, που έχει ακόμη πολλές πρόοδους να σημειώσει. Μπορούμε να κάνουμε μια ορθή μεταφορά χωρίς να εγκρίνουμε οριζόντια νομοθεσία, αλλά συμπεριλαμβάνοντας οι βασικές αρχές σε τομεακή νομοθεσία. Αυτή είναι μια τεχνική προσέγγιση, η οποία καμιά φορά είναι δύσκολη και πελέγει, για παράδειγμα, στη Γερμανία και στη Γαλλία. Κάτι σαφές βέβαια είναι ότι η οριζόντια νομοθεσία δεν επαρκεί. Το η εργασία είναι πολύ ε, μεγαλύτερη όσον αφορά την προσαρμογή της ε, υφιστάμενης νομοθεσίας. Έχουν ήδη ε, γίνει κάποιες τροποποιήσεις ή έχουν ξεκινήσει τροποποιήσεις σε κάποια κράτη-μέλη. Και για να σας δώσω μια ιδέα, πάνω από 600 από 600 νομοθετικές πράξεις ε, έχουν μέχρι σήμερα ε, τροποποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν καθυστερήσει στην προετοιμασία της ε, τροποποίησης της νομοθεσίας τους. Αυτή είναι ακριβώς τη δουλειά έχω σκοπό να κάνω στις επισκέψεις μου στις διάφορες πρωτεύουσε. Δεύτερο, ενιαία θηρίδα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει στην πράξη η οδηγία να ε, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του ο κάθε πολίτης ε, σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενιαία θηίδα ισχύει σε 21 κράτη-μέλη, σε 6 όχι. Και επομένως ε, μπορεί να σημειωθεί ακόμη κάποια πρόοδος. Ε, σε μερικές περιπτώσεις ε, δεν γίνονται ε, συναλλαγές, για να το πούμε έτσι, στο πλαίσιο της ενιαίας διείδας. Είναι απλώς ενημερωτική, ενημερωτικός ο ρόλος τους και πρέπει να ολοκληρωθεί η λειτουργία τους για να μπορούν να είναι συμβατές οι θηρίδες αυτές με την λειτουργία που προβλέπει η οδηγία. Πρόκειται για τις πύλες, τους μοχλούς για την επίτευξη της εφαρμογής της οδηγίας. Όσον αφορά τώρα την διοικητική συνεργασία και εδώ υπήρξαν κάποιες πρόοδοι ε, στο πλαίσιο των δικτύων διοικητικής συνεργασίας και για τη διευκόλυνσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίδρυσε το ηλεκτρονικό σύστημα διοικητικής συνεργασίας που είναι πολύγλωσσο πολλές αρμόδιες υπηρεσίες, 4.500 περίπου, από όλα τα κράτη-μέλη έχουν καταχωρηθεί στο συγκεκριμένο σύστημα πληροφοριών και πάνω από 1.300, πάνω από 1.300 ε, ανταλλαγές πληροφοριών έγιναν το, 1000, το 2009 και έδωσαν τη δυνατότητα να δοκιμαστεί το σύστημα. Αυτό σημαίνει τεράστιο δυναμικό, όπως το καταλαβαίνετε. Υπάρχει το σύστημα IMI, το ε, σύστημα πληροφοριών της εσωτερικής ε, αγοράς και θα συνεχίσουμε βέβαια τις προσπάθειές μας για την καλύτερη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Ενδεχομένως να ήταν χρήσιμο να ακούσουμε ε, την κυρία Γκέπχαρντ ε, και τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής σας για τα καταληκτικά σχόλια. Υπάρχουν πρόοδοι, αλλά δεν είναι επαρκείς. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν μείνει πίσω και πρέπει να διπλασιάσουν την προσπάθειά τους. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός ως προς αυτό. Και πρέπει να πω ότι θέλω να δώσω κάποιο χρόνο, αλλά όχι αόριστο χρόνο. Δεν είναι δυνατόν, επαόριστον δηλαδή, να καθυστερεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πρέπει με το συντονισμό να καταλήξουμε στην εφαρμογή όλων των εργαλείων που, έχουν, που συνδέονται με την οδηγία αυτή και ελπίζω όλοι σας να ακούτε αυτή την έκκληση στην ευθύνη που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια, εκτός από το κομμάτι το νομοθετικό που τους ενδιαφέρει για τη μεταφορά του εθνικού δικαίου, για την προσαρμογή ε, της εθνικής νομοθεσίας, ε, τα εθνικά κοινοβούλια συμπεριλαμβάνουν πολιτικούς των οποίων η ε, πειθό και η σκληρή δουλειά θα βοηθήσει ε, την ε, καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας ε, στην χώρα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει και εκείνη τις δικές της ευθύνες. Η προθεσμία της εφαρμογής δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Η ενιαία θηρίδα θα παραμείνει πολύ σημαντική μακροπρόθεσμα. Και θέλω να αναπτύξουμε επίση, γιατί το χρειαζόμαστε πολύ συχνά, όχι, σε πολύ σημαντικό βαθμό, όχι μόνο την οδηγία, αλλά και τα συστήματα πληροφόρηση στα αμοιβαία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό επίση σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και εγώ θα είμαι διαθέσιμος για να συμμετέχω στις συναντήσεις σας και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα σας δω και στις πρωτεύουσές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε στην κριτική επικοδομητική αξιολόγηση της ε, ε, οδηγία για τις υπηρεσίες, που είναι τόσο σημαντική για την εσωτερική αγορά και τη λειτουργία, σας, τη λειτουργία της. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο θα φτάσουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Θα ήθελα κυρία Γκέπχαρτ να μας συνοψίσει την κατάσταση. Είμαστε όμως ιδιαίτερα ευγνώμονες κύριε Επίτροπε που ε, προσήλθατε εδώ και είμαι σίγουρος ότι ότι ορισμένα μέλη εθνικών κοινοβουλίων που δεν έχετε επισκεφθεί ακόμα ε, θα ε, χαρούν ιδιαίτερα που σας βλέπουν. Βεβαίως είστε πολύ δραστήριος και μεταβαίνετε από χώρα σε χώρα, αλλά ίσως ε, δεν έχετε μεταβεί σε όλες. Η κυρία Ντεκράς μετά την... Μάλλον ο κύριος θα μας πει για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και θα αναλάβετε και μετά την... Ε, θα, θα αναλάβετε και την Προεδρία μετά την Ισπανική. Ναι, ε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαρνιέ, ο οποίος ε, βρίσκεται εδώ. Μας χαροποιεί αυτό ιδιαίτερα και βλέπουμε την ανάγκη ύπαρξης αυτής της οδηγίας, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προοπτική αυτής της οδηγίας, ποια, ποιο είναι το ευεργέτημα που απορρέει από μια τέτοια οδηγία, την αύξηση εμπορικών δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών. Και αυτό έχει αντίκτυπο και στην απασχόληση η αρχική, μεταξύ της αρχικής οδηγίας του 2002 και της παρούσας, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και η συγγήτρια τόνισε ότι δεν πρέπει πια να μιλάμε για την οδία Μπόλκενστάιν. Πρόκειται για κάτι το εντελώς διαφορετικό. Άρα η ο ευεργετικός αντίκτυπος θα είναι διαφορετικός μεταξύ της πρώτης έκδοσης Μπόλκενστάιν και της βελτιωμένης έκδοσης και πώς θα φτάσετε σε μια εξισορρόπηση των διαφόρων ε, επιχειρημάτων εάν υπάρχει μια δυναμική πορεία προς το μέλλον. Από πότε έχουμε αυτά τα στοιχεία αξιολόγησης από τα 60 στα 140 ε, δισεκατομμύρια από το 1 στο 1,5 δίκτυα ανάπτυξης, αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται για μια έκδοση η οποία δεν είναι επίκαιρη. Θα το επιβεβαιώσω, διότι αν ε, μου δίδονται αυτά τα στοιχεία σήμερα από την υπηρεσία μου, θα πρέπει να, έχουν, να είναι μια τάξη μεγέθους τα αριθμητικά αυτά τα, τα στοιχεία ορίζονται από το κείμενο στην τελική μορφή την όρισε το Κοινοβούλιο και όχι με βάση την αρχική έκδοση Μπόλκενστάιν. Merci, très εντάχει γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ που παρίσταστε εδώ ε, κύριε Πίτροπε. Μιλήσαμε για πληροφόρηση προς τους πολίτες, διότι γνωρίζει ο πολίτης ότι υπάρχουν πολλά ψευδή στοιχεία που αναφέρθηκαν για αυτή την οδηγία. Και αυτό αφορά και τους πολιτικούς. Νομίζω λοιπόν όταν ε, οριοθετήσουμε το πεδίο εφαρμογής και όταν οι ενιαίες ε, θηρίδες είναι αποτελεσματικές, γιατί μιλήσαμε για τον πολυσχηδή χαρακτήρα μεταφοράς αυτής της οδηγίας, αυτό που έχει σημασία είναι οι πολίτες να ευεργετηθούν ε, οικονομικά και κοινωνικά με βάση την κυκλοφορία αυτών των προϊόντων. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν η υπόψη από τον πολίτη κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα μεγάλα εθνικά μέσα θα πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες κάθε κράτους με τη συνεργασία των κοινοβουλίων για να εξηγήσουμε στα μέσα ενημέρωση ότι πρέπει να επεξηγήσουν αυτό το πλαίσιο και τι είναι θετικό για την καθημερινή ζωή του πολίτη. Έτσι μόνο θα βελτιωθεί η Ευρώπη. Και σας ευχαριστώ γιατί το υπογραμμίσατε αυτό. Good. Uh, Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Ο κύριος Πεντικά από το, την Ιταλική Γερουσία και ο κύριος Κόσουσνικ στη συνέχεια. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κάποιος άλλος. Μετά ο κύριος Μπαρνιέ θα μπορέσει να συνοψίσει. Ο κύριος Πέντικα έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Μία ερώτηση θα ήθελα να υποβάλω. Ε, όταν περνάει ένα προεδρικό διάταγμα όπως έγινε σε εμάς που αντιτίθεται στην οδηγία περιπηρεσιών, πώς μπορούμε να αντιταχθούμε σε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να πω ότι οι εξαιρέσεις είναι το πιο λεπτό θέμα που αφορά την οδηγία διότι γίνεται μάλλον δίνεται μία εκτατική ερμηνεία της οδηγίας έτσι ώστε να μην είμαστε σίγουροι τι καλύπτουμε με τις παροχές αυτές και με τον ενιαίο πάροχο. Στη μεταφορά που έγινε από την Ιταλία με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης εβδομάδας φαίνεται ότι το καθεστώς των εξαιρέσεων χρησιμοποιήθηκε ε, υπερβαίνοντας το πλαίσιο των ε, Βρυξελών. Το άρθρο 2 του διατάγματος προβλέπει εξαιρέσεις όταν μιλάμε για δέκο και υπηρεσίες κοινού ενδιαφέροντος που επιλέγονται και δρούν μέσα στα πλαίσια ε, μιας υπηρεσίας που παρέχει ένα νομικό πρόσωπο. Γι' αυτό νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιφάσκουμε με την αιτιολογική σκέψη παριθμό 17 της οδηγίας, όπου λέει ότι η ΔΕΚΟ είναι υπηρεσίες που καλύπτουν ένα οικονομικό πλαίσιο δυνάμει της παρούσης οδηγίας και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αντιτασσόμαστε στην οδηγία διότι στην περίπτωση του φυσικού αερίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας μιλάμε για υπηρεσίες ε, εθνικού οικονομικού συμφέροντος. Γι' αυτό φαίνεται ότι η Ευρωπαίος συμφεροντος γι αυτο φαινεται οτι ο ευρωπαιος νομοθετης δεν ήθελε να αποκλείσει τις ΔΕΚΟ και η Ιταλική κυβέρνηση προέβη και δέχτηκε εξαιρέσεις που δεν είναι αποδεκτές. Θα πρέπει λοιπόν να μας ξαναπασχολήσει αυτό το θέμα για να δούμε κατά πόσο φτάσαμε στους απότερους στόχους της οδηγίας, έτσι ώστε να καλύπτουμε και τις δέκο γενικότερα για να μπορέσει να πραγματοθεί η ενιαία αγορά. Μια άλλη σκέψη. Θα θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Εμείς είμαστε κόμμα της αντιπολίτευσης και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επιβάλλουμε τους κανόνες των Βρυξελών και κατά πόσο η κυβέρνηση δεν θα ήταν σκόπιμο στο προεδρικό διάταγμα να προέβαινε σε μία κατεξουσιοδότηση πράξη για την κοινωνική προστασία των πολιτών μέσα στα πλαίσια των διασυνοριακών υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τους πιο αδύναμους εργαζόμενους και να μην ε, καλύπτουμε μόνο τις ε, ιδιωτικές μεγάλες επιχειρήσεις όπως ισχύει στον τομέα της αποχέτευσης και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κάτι το οποίο δεν θα βελτιώσει την ίδια την παροχή της ποιοτική υπηρεσίας. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν κατά πόσο καλύπτουμε, καλυπτόμαστε σωστά πίσω από την ε, οδηγία αυτή. I'm, του χρόνου της Κομισιόν και ήταν και μακροσκελής η παρέμβασή σας, οπότε δεν νομίζω ότι μπορείτε να περιμένετε από τον Επίτροπο να απαντήσει σε όλα, έτσι. Να πω όμως στους αδέλφους από το Κοινοβούλιο ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα είναι αύριο το πρωί εδώ στις 9 για να μας μιλήσει για το πρόγραμμά του. Οπότε μην αγχώνεστε και αύριο το πρωί έχετε χρόνο να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Οπότε ας κλείσουμε τώρα την, τις Α μην πάρουμε μάλλον άλλε ερωτήσει. Ο κύριο Μπαρνιέ μπορεί να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια. Μετά θα πάρει το λόγο η κυρία Και εγώ θα κλείσω την συνεδρίαση και ελπίζω να είμαστε και εντό των χρονικών ορίων μα. Κύριε Επιτροπέ, παρακαλώ, κάποια καταληκτικά σχόλια. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι εδώ σήμερα και θα έρθω και αύριο το πρωί, μήπως να κοιμηθώ εδώ. Καλή ιδέα μου ακούγεται. Σχόλιο εκτό μικροφώνου. Λέει ο κύριος, Χάρμπουρ, έχουμε και πολλές προσκλήσεις σε δείπνο αν θέλετε. Τέλος πάντων, να σας ε, σοβαρευτούμε λιγάκι. Ήθελα απλώς να επιβεβαιώσω αυτό που είπα προηγουμένως. Ε, οι συνεργάτες μου μου λένε ότι όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο που ανέφερα προηγουμένως, ε, τα ε, στοιχεία που σας ανέφερα, κατά προσέγγιση βέβαια, είναι του 2007. Από μία ανεξάρτητη μελέτη από το CPB. Έτσι λεγόταν ε, η εταιρεία που το είχε αναλάβει και υπήρξε και μία προοπτική στο πλαίσιο της έρευνας αυτής ε, και αυτά ακριβώς τα στοιχεία είναι που σας έδωσα κατά προσέγγιση. Ο κύριος Πέντικα είπε πολλά πράγματα για τα οποία, στα οποία δεν θα απαντήσω σε πολύ λεπτομερώς. Τον άκουσα όμως με πολύ προσοχή σε πολλές περιπτώσεις. Η Γαλλία για παράδειγμα έχει εξαιρέσει κάποια κοινωνικά θέματα όπως για παράδειγμα ε, τους ε, βρεφονιπιακούς σταθμούς. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα συμβιβασμό που είχε ω αποτέλεσμα κάποια κοινωνικά, κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες να μείνουν εκτός, αλλά όχι όλες. Αυτές που παρήχε το κράτος, ε, οι συμβεβλημένοι φορείς με το κράτος, ε, εξαιρέθηκαν. Αντιθέτως, οι ιδιωτικές είναι, διέπονται από την οδηγία. Κοιτάξτε, Κάποιες χώρες αυτό το μετέφεραν και στην εθνική τους νομοθεσία. Ανησυχώ και εγώ, όπως και οι εθνικοί βουλευτές και οι ευρωβουλευτές, για το θέμα της προστασίας ε, των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κοινή ωφελία. Πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον πώς θα γίνει αυτή η προστασία, πώς θα εξασφαλίσουμε νομικώς κάτι τέτοιο μέσω μια οδηγίας πλαίσιο, ε, τι νομικό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξει, κάποιε κάποιες οδηγίε. οδηγίες. Κοιτάξτε, δεν είναι τίποτε γραμμένο στην πέτρα, εγώ ανοιχτό είμαι και θα το συζητήσουμε και αύριο το πρωί. Πρόκειται για υπηρεσίε ε, που πραγματικά επηρεάζουν πολύ τους πολίτες. Και βεβαίως πρέπει και να προστατευθούν και να εξασφαλιστούν και δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις αποδυναμώσει αυτές τις υπηρεσίες που είναι τόσο υποφελείς για τους πολίτες. Και κάτι ακόμη, για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, το λέω και στα Εθνικά Κοινοβούλια, αν έχετε ερωτήσεις ε, που δεν τις θέσατε ή αν δεν είναι επαρκής οι απαντήσεις μας, ε, μπορούμε και με email να ε, συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεών μας ε, ή στις επισκέψεις στις χώρες, στις χώρες σας. Βέβαια, στο Λονδίνο έχω πάει ήδη πολλέ φορέ και πήγα και πριν μερικέ εβδομάδε. Πρέπει να πάω και στι υπόλοιπε πρωτεύουσε. Κυρία Βερνιό, κάνατε μια ερώτηση που είναι πολύ σημαντική και κάνατε και πολύ σημαντικές προτάσεις όσον αφορά την ε, κατάρτιση των πολιτών. Όταν τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει κάποια από τα μέσα της για να κάνει εκστρατείε ε, και κάνει ήδη κάποιες, ειδικότερα για να έρθει σε επαφή με τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή, να τους προσεγγίσει στην καθημερινή τους ζωή με πράγματα που είναι εποφελείς για τους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Μιλούσαμε για την οδηγία Μπόλκενστάιν, τη συγκεκριμένη εκστρατεία στη χώρα μου, αυτή η υπόθεση με τον Πολωνό Ιδραυλικό. τα θυμάστε. Εγώ έμαθα το μάθημά μου και θα το λάβω πολύ σοβαρά υπόψη ως Ευρωπαίος Επίτροπος αποφάσισα ότι όλα τα επόμενα κείμενα που θα παρουσιάσω εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν είναι λογικά και σημαντικά και έχουν αντίκτυπο σε κάθε μία από τις χώρες, μαζί τη στιγμή που γίνεται μία πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών, όταν λοιπόν θα κάνει την πρόταση της ε, και στα Εθνικά Κοινοβούλια και στους Ευρωβουλευτές ε, θα διαθέτει μέσα ενημέρωσης ε, είτε CD είτε έγγραφα στις γλώσσες τους και θα δείτε στη διάθεσή σας στις περιφέρειές σας για να μπορείτε να ξεκινήσετε μία συζήτηση. Αυτό ήταν το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας και εγώ αποφάσισα να το κάνω στην πράξη. Θα ήθελα να το κάνω και νωρίτερα, γιατί πραγματικά μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το χάσμα, αυτή η έλλειψη σχέση μεταξύ της συζήτηση στις Βρυξέλλες και στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Για τα σημαντικά λοιπόν θέματα που θα προτείνω, και για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για την παγίωση ε, της εσωτερικής αγοράς και για το θέμα της ε, ρύθμισης της ε, εποπτείας, ε, όχι κάθε εβδομάδα, όχι για κάθε κείμενο, αλλά για τα σημαντικά κείμενα θα διαθέσω και στα εθνικά κοινοβούλια, σε κάθε μία από τις 27 χώρες, στη γλώσσα τους, αλλά και στους ευρωβουλευτές υλικό, ενημερωτικό για να μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση γύρω από εσά, να είναι γνωστές, να γνωστοποιήσετε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μπορείτε μετά στη συνέχεια να ε, μεταφέρετε εσείς ε, σε εμά τις προτάσεις ε, ή την, τις απόψεις των πολιτών. Αυτά ήθελα να πω. Ούτως ή άλλως αυτή η αλλως αυτη η ενημερωση των πολιτών είναι κάτι που πραγματικά με απασχολεί πάρα πολύ και με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ και για την προσφορά σας και για τη διαθεσιμότητα που δείχνετε και εμείς την εκτιμούμε, φαντάζομαι και τα εθνικά κοινοβούλια. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή με τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Και όπως σας είπα και πιο πριν, η Εύελιν θα, πάρει τώρα, θα είναι η συγκήτρια για την έκθεση για την μεταβατική έκθεση και φαντάζομαι ότι θα έρθει σε επαφή μαζί σας. Εύελιν, σου δίνω λίγα λεπτά για να κλείσεις και μετά να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που έκαναν τον κόπο να έρθουν εδώ στις Βρυξέλλες και να συζητήσουν μαζί μας για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμος ο διάλογος αυτός. Εγώ έλαβα πάρα πολύ χρήσιμες, πολλές πληροφορίες. Δεν μπορώ να μπω στη λεπτομέρεια όλων γιατί θα λαπανούσα πολύ χρόνο. Αλλά θα ήθελα να κάποια σχόλια να τα κάνω. Που είναι σημαντικά. Καταρχήν, αυτή η συνεργασία που βρίσκεται στο πνεύμα και στο γράμμα της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας, της συνθήκης της Λισαβόνας μάλλον. Είναι, μάλλον, είναι πολύ πιο ενισχυμένη τώρα με τη συμμετοχή και τη συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Βέβαια πάμε και λίγο παρακάτω από την συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά στην κατεύθυνση που, για την οποία μίλησε και ο Επίτροπος Μπαρνιέ. Ότι δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σύνδεση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή συζήτησης και των εθνικών συζητήσεων που τρέχουν. Αυτό σημαίνει ότι συζητούμε και μεταξύ μα. Και ξέρουμε περί τίνο συζητούμε. Ganz wichtige Sache. Der zweite Punkt, der herausgegangen ist aus den vielen Diskussionen, die wir hatten, ist, dass wir ein είναι σημαντικό επίση να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη των πολιτών, να μπορούν δηλαδή να νιώθουν ε, οικία στην Ευρώπη στην οποία ζουν να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά του για την προστασία του ω καταναλωτέ, για, για τα εργασιακά του δικαιώματα. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά. Και επίση έχουμε και τη συμβολή τη κυρία Γιάνσεν, πολύ σημαντική συμβολή τη, γιατί έτσι πρέπει να συζητήσουμε άλλη μια φορά πώς μπορούμε ε, πώς μπορούν να, συγκεραστούν όλες αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οδηγίες για τις αποσπάσεις. Ε, έχει δημιουργήσει και αυτή πολλά προβλήματα στη Σουηδία με τις ιδιαίτερες συνθήκες τις συμβασιακές που θέτει για τα, για τα συνδικάτα. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα συζητήσουμε. έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις διόδους συνεργασίες που έχουμε, συνεργασίας που έχουμε και να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Γιατί σε κάποια προβλήματα που υπάρχουν μάλλον τα, κάποια ε, προβλήματα που υπάρχουν μπορούν να λυθούν όχι μέσω τη οδηγία για τις υπηρεσίε, αλλά μέσω άλλων νομοθετικών πράξεων, δηλαδή από των άλλων νομοθετικών τομέων. Επίσης, η εθνική, τα κέντρα εξυπηρέτηση, οι εθνικοί συνομιλητέ, είναι σημαντικά γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι της οδηγίας για το άνοιγμα των αγορών στην εσωτερική αγορά, στην κοινή αγορά που έχουμε και την οποία φροντίζουμε έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να κινούνται και να παρέχουν, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ευρώπη. Είτε είναι πάροχοι υπηρεσιών, είτε θέλουν να εγκατασταθούν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Να μπορέσουμε να τους διευκολύνουμε. Και αυτό είναι πάντα ένα σημείο για το οποίο μιλά ο Επίτροπος Μπαρνιέ, για την ενημέρωση. Το συζητήσαμε και με του εκπρόσωπου τη τους της Κομισιόν που είναι ήδη εδώ. Είπαμε ότι θα ήταν απαραίτητο να υπάρξει μια ενημερωτική εκστρατεία για τι υπηρεσίε και κυρίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Να ε, τους ενημερώσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι συνομιλητέ, γιατί έχουμε διασπιστώσει σε πολλέ συζητήσει που κάνουμε ότι πολλοί που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από όλο αυτό δεν ξέρουν ότι καν υπάρχει αυτό το ενιαίο κέντρο ε, ε, Οπότε καλό θα ήταν όλες αυτές οι πληροφορίες να δοθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς και ε, υπάρχει αυτό το λογότυπο το οποίο βγήκε. Μια αρχή είναι και αυτό. Ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι και το κίνητρο για την ενημερωτική αυτή καμπάνια. Νομίζω ότι και αυτό είναι αρκετά σημαντικό στην ε, συζήτηση που κάναμε σήμερα. Κλείνοντας και σε σχέση... Κλείνω, κλείνω πρόεδρε και σε σχέση με το σημείο της, ε, του πεδίου εφαρμογή τη Οδηγία για τις υπηρεσίες. Ακόμη υπάρχει ανάγκη για συζήτηση, είναι σαφές αυτό, υπάρχει ανάγκη για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Την εντύπωση αυτή είχα και εγώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που είπε ο Επίτροπος τώρα στο τέλος και το οποίο πάντα παίζει ρόλο στις συζητήσει για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Είπαμε ότι θα, κλείσουμε τις, θα αποκλείσουμε τις υπηρεσίες κοινή οικονομικής ωφέλειας. Δεν θέλαμε να πούμε ότι δεν θα φροντίσουμε να κάνουμε τίποτα για αυτές τις υπηρεσίες. Είπαμε απλώς ότι δεν θα, εμπίπτουν σε αυτή την οδηγία και ότι θα έχουμε ένα, ένα δίκαιο πλαίσιο για αυτές, τις, α, για αυτές τις ειδικές ε, υπηρεσίες. Και ακόμα βέβαια δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Με ποιο τρόπο θα λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Αλλά ένα είναι σαφέ ότι δεν θα αφήσουμε τα πράγματα έτσι όπω είναι και θα πούμε απλώ τα κράτη-μέλη α πράξουν αναλόγω ή α πάνε στο δικαστήριο να πάρουν την ομολογία να δούνε τι λέει. Ε, πρέπει να δώσουμε ένα ερώ... ένα μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα το διαχειριστούμε το θέμα αυτό, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι και ένα από τα αποτελέσματα, τι συνέπειε που πρέπει να δούμε πώ θα επηρεάσουν. Ναι, ε, το ξέρω, θα τελειώσω, θα τελειώσω, θα σου κάνω τη χάρη πρόεδρε, τελειώνω τώρα. Η ομάδα μου ακόμη δεν έχει καθορίσει ποιος θα αναλάβει την γνωμοδότηση. Έχουμε μια δημοκρατική διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσει η ομάδα μου να είμαι εγώ η συγκήτρια ώστε να μπορέσω κι εγώ να συμβάλλω στην, στην γνωμοδότηση με όλα αυτά τα σημεία τα οποία τώρα μου απαγορεύει ο πρόεδρος να πω. Λόγω χρόνου βέβαια. I think your would be, um, Νομίζω ότι ε, θα είχαμε χάσει μια πολύ ε, ωραία ευκαιρία αν δεν σου δίναμε τη δυνατότητα να είσαι εισηγήτρια και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν. Κυρίες και κύριοι, ήταν μεγάλη μας ε, χαρά να σας έχουμε εδώ μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ που καταβάλατε την προσπάθεια να έρθετε εδώ. Ελπίζω η συνεργασία να είναι συνεχής ο Επίτροπος χρησιμοποίησε μία φράση. Όταν μίλησε για τις ενιαίες θηρίες, μίλησε σαν να ε, δίνουμε ζωή στις υπηρεσίες. Αυτή είναι και η ουσία, γιατί έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς ένα μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου ε, παίρνει ζωή στη χώρα σας και κινείται προς την πραγματική αγορά. Και ό,τι ε, και να πείτε για τον Πολωνό υδραυλικό, θυμάμαι ότι η κυρία Χάνσλεϊ είχε φέρει έναν υδραυλικό Πολωνό εδώ στο Κοινοβούλιο, ήταν πολύ όμορφος, πάρα πολύ όμορφος. Και θυμάμαι ότι όταν πήγα στο Κέντορσε στο Υπουργείο Εξωτερικών πριν δώσουμε τελική μορφή στη δεξίωση είδα την αφίσα του Πολωνού Ιδραυλικού εκεί στο Σε. Και αυτό έδειχνε ότι θα δώσουμε ζωή πραγματικά σε αυτή την ε, οδηγία. Θέλουμε κάτι εξίσου εικονικό και γραφικό. Ελπίζω μας βοηθήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και θα συνεδριάσουμε ως Επιτροπή αύριο στις 9 το πρωί στο 1G3 όπου θα έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο και πάλι. Στις 10 και 4 έχουμε ψηφοφορίες. Μην ξεχάσετε την ηλεκτρονική σας κάρτα και χαίρετε.